Colleghi, collega Lunacek. Συνάδελφε, Λούνατσεκ, ησυχία. Ε, ricordo... Σας υπενθυμίζω τις αλλαγές που έγιναν στην ημερήσια διάταξη της αυριανής μας συνεδρίασης για τις 13 Ιουλίου δηλαδή αντί για την ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Αχμέτ Νταβούτογλου, που προβλέπεται προβλεπόταν allora colleghi Αγαπητοί συνάδελφοι, σας υπενθυμίζω τις αλλαγές στην αυριανή ημερήσια διάταξη 13 Ιουλίου. Στη θέση της ανταλλαγής απόψεων με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Αχμέτ Νταβούτογλου, προβλέπεται στις 4 και 4 μέχρι τις 5.30 μία συνάντηση με τον Μαχμούτ Τζιμπρίλ, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου, ε, σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη. Και έχουμε και ανταλλαγή απόψεων, μάλλον δεν θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον Μπερναρντίνο Λεόν, οριστέντα ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής ε, Ένωση στη Νότια Μεσόγειο, γιατί ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί ο διορισμός του. Άρα να βάλετε αυτή η ανταλλαγή απόψεων για μετά το καλοκαίρι. Περνάμε λοιπόν στο ε, τρίτο θέμα που είναι η εκλογή ενός νέου αντιπρόεδρου. Σας υπενθυμίζω ότι μετά την παρέτηση του Ντομινίκ Μπομπί, ως ε, τρίτος αντιπρόεδρος προτείνεται ο Τόκια Σαΐφη. Η, η. κυρία Τόκια Σαΐφη είναι η μόνη υποψήφια για την θέση του τρίτου ή της τρίτης αντιπροέδρου. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν αντιρρήσεις, προβλέπω εκλογή διαβοής. Bene, allora vista l'unanimità dei consenti dei consenti θα ήθελα λοιπόν να προσέλθετε εδώ στη, στα έδρανα του Προεδρείου. Congratulations. Je me félicite. Αρχίζουμε με την δημόσια ακρόασή μας σε σχέση με την εξωτερική πολιτική της ε- Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις χώρες BRICS και άλλες αναδυόμενες δυνάμεις. Ποιοι είναι οι στόχοι και οι στρατηγικές. Θα ήθελα τα μέλη του πάνελ να έρθουν εδώ. Η κρίση της Λιβύης και η πρόσφατη συνάντηση των εκπροσώπων των χωρών ε, BRICS στην Κίνα καταδεικνύει ότι οι χώρες αυτές είναι πολύ σημαντικές και από πολιτικής ε, πλευράς και από οικονομικής. Εάν σκεφτούμε την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις ε, χώρες αυτές και τις άλλες αναδυόμενες δυνάμεις βλέπουμε ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν ε, αυτές οι σχέσεις. Μετά από έκθεση μετά από την έκθεση πρωτοβουλίας του κύριου Σάριους Βόλσκι προτάθηκε αυτή η ακρόαση. Δυστυχώς ο κύριος Σάριους Βόλσκι είναι άρρωστος και θα πρέπει να προχωρήσουμε στην ακρόαση εν τη απουσία του. Ζήτησε όμως από τη γραμματεία να ε, μπορέσει να καταγράψει τις παρεμβάσεις για να τις συμβουλευτεί. Έχουμε πέντε ομιλητές. Καταρχήν τον Αλφρέτο Βαλιαντάου, εκ δεξιών του Προέδρου, που είναι ε, πρόεδρος ε, της Μερκοσούρ, της ε, ε, της έδρας της Μερκοσύρ στο Ινστιτούτο Πολιτικών Μελετών του Παρισιού. Ε, τον Ενρίκε Μόρα Μπεναβέντε, τον Άντρου Σμόλ. Ενρίκε Μόρα Μπεναβέντε, ε, λοιπόν, που είναι ε, διευθυντής της ε, πολιτικής εξωτερικών υποθέσεων της Ισπανίας, Σίριλ Ναν, ο οποίος είναι υπεύθυνος των ασιατικών υποθέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων Εξωτερικών της Γερμανίας και στη συνέχεια τον κύριο ε, Βιορέλ Μπουντούρα, ο οποίος είναι υπεύθυνο της ΕΙΕΔ σε σχέση με την κατάσταση στην Ασία. Θα ακούσουμε λοιπόν τους πέντε εισηγητές μας και Καταρχήν θα ακούσουμε τους δύο πρώτους, θα δώσουμε το λόγο στους βουλευτές για σχόλια ή ερωτήσεις και μετά τους υπόλοιπους τρεις και θα δώσουμε το λόγο στους βουλευτές για ενδεχόμενες ερωτήσεις. Σήμερα η ημερήσια διάταξη προβλέπει και μία ανταλλαγή απόψεων ε, με τον κύριο Νουζαΐφη, εκπρόσωπο τύπου του Συμβουλίου Αντιπροσώπων του Ιράκ. Κατά τις 5.30 θα πρέπει λοιπόν να λήξει η δημόσια ακρόαση μέχρι τις 5.30. Δίνω το λόγο στον κύριο Βαλιαντάου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή θα μιλήσω στα αγγλικά γιατί νομίζω ότι είναι καλύτερα. Είμαι ε, ε βραζιλιάνος, άρα είμαι το B των BRIC. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι ε, οι χώρες BRIC δεν είναι μια πολιτική κατηγορία, αλλά μια στρατηγική επένδυση που την ε, εφήβρε η Goldman Sachs πριν από καμιά δεκαετία χρόνια. Τα μέλη της ε, ομάδας αυτής, με πρωτοπόρα τη Βραζιλία, προσπαθούν να δημιουργήσουν μια πολιτική οντότητα, συμπεριλαμβάνοντας και την Νότιο Αφρική. Ε, στο πλαίσιο της πολιτικής ορθότητας. Η αλήθεια όμως είναι ότι τα BRICS αυτή τη στιγμή είναι μια βιτρίνα που δεν, ε, δεν έχουν ένα κοινό όραμα, ούτε μια κοινή στρατηγική, ούτε καν μια κοινή αμυντική στάση. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι κάθε μία από τις χώρες BRICS ε, δεν ενισχύει το ρόλο της και τη θέση της. Αντιθέτως, θα ήθελα όμως να αφήσουμε εκτός τον BRICS τη Ρωσία γιατί ε, δεν είναι αναδιόμενη δύναμη, είναι αναδιόμενη υπερδύναμη. Συνεπώς ας μιλήσουμε για τις υπόλοιπε χώρες. Ε, Βραζιλία, Κίνα, Ινδία ε, έχουν μια ισχύ η οποία είναι αποτέλεσμα της οικονομικής τους ισχύω. Η οικονομική ισχύ όμως φέρνει και πολιτική και στρατιωτική ισχύ και όλες αυτές οι χώρες ε, αυξάνουν τους, τις αγορές και τους στρατιωτικούς προϋπολογισμούς, τις αγορές ε, πολεμικού υλικού ε, και ενισχύουν τη θέση τους στα διεθνή φόρα. Αρχίζουν λοιπόν να επηρεάζουν ε, την κατάσταση σε πολλά στρατηγικά θέματα όπως ε, τροφιμική ασφάλεια, ενεργειακή ασφάλεια, ασφάλεια στις θάλασσιες μεταφορές, περιφερειακή ασφάλεια, ε, ανθρωπιστική δράση, διατήρηση ειρήνης, κλιματικές αλλαγές, λειτουργία του ΟΗΕ και άλλων διεθνών οργανισμών κλπ. Η πρωτοβουλία Βραζιλίας-Τουρκίας, ε, για παράδειγμα, για το, ε, για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ήταν αποτυχία. Αλλά έδειξε ότι αυτές οι χώρες έχουν τη βούληση να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους μεγάλα ζητήματα. Όλοι γνωρίζουμε πως ε, στο μέλλον θα είναι όλο και πιο δύσκολο να εξασφαλίζουμε πολυμερείς συνενέσεις για τα μεγάλα παγκόσμια προβλήματα χωρίς, ε, θα είναι δύσκολο να εξασφαλίζουμε τέτοιες συνενέσεις χωρίς τη συμμετοχή των χωρών αυτών. Και αυτή είναι και η λογική του G20, να τις βάλουν στο παιχνίδι. Η μεγάλη δυσκολία είναι ότι οι χώρες αυτές ε, δεν, είναι δεν αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα. Ανάλογα με το ποιο θέμα συζητείτε, μπορεί να έχουν τελείως αντιδιαμετρικές απόψεις. Για παράδειγμα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η Ρωσία και η Κίνα δεν συντάσσονται πάντοτε με τη Βραζιλία και την Ινδία. Μπορούμε τη στάση τους να, σε ό,τι αφορά τη διεθνή παγκόσμια τάξη να την ορίσουμε ως ε, ε, ε, ε, ε κερδοσκοπική πολυμερή στάση. Ε, θέλουν περισσότερη ισχύ, χωρίς όμως ε, απαραίτητα να θέλουν να ε, χρηματοδοτούν αυτή την διεύρυνση του πολυμερούς χαρακτήρα των διεθνών οργάνων. Θέλουν δηλαδή να έχουν μια, στάση, μια δυνατότητα βέτο, χωρίς όμως να είναι πολύ ε, συμμετοχικές σε, αυτές, σε αυτούς τους ε, φορείς, σε τους διεθνείς οργανισμούς. Συνεπώς, ε, έχουν μεγάλες ευθύνες στη διατήρηση της οικονομικής, παγκόσμιας οικονομικής τάξης και αυτό τις φέρνει πιο κοντά στις ΗΠΑ από ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε όλα τα θέματα σχετικά με τη ρύθμιση παγκόσμια οικονομίας και του παγκόσμιου συστήματος. Αυτό αυτό όμως σημαίνει ταυτόχρονα ότι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό και από την, πολύ, ε, από την καλή λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας και της παγκόσμιας τάξης. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε από μόνες τους αντιπροσωπεύουν το 1 τρίτο της ιδιωτικής κατανάλωσης του κόσμου. Η Ευρώπη το άλλο τρίτο, η Κίνα το 3% Οπότε αν η Κίνα δεν μπορεί να εξάγει στις ΗΠΑ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα πληγεί και η οικονομική της ισχύ. Η ανάπτυξη όμως κατά βάση προέρχεται από αυτές τις χώρες. Οπότε οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από αυτές τις χώρες. Συνεπώς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση αλλοεξάρτησης. Και αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ε, άλλη διέξοδος από το να πάρουμε στα σοβαρά αυτούς τους καινούριου παίκτες και να τους συμπεριλάβουμε. Ένα παράδειγμα πρόσφατο πρόβλημα που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Κίνα. Ε, φόροι του άνθρακα επί των αεροπορικών εταιριών που οι Κινέζοι είπαν ότι αν κάνετε κάτι τέτοιο δεν θα ξαναγοράσουμε Airbus. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αρχίζουν και λένε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν θέλετε να ρυθμίζετε ε, την οικονομία θα πρέπει να μας λαμβάνετε υπόψη. Οπότε οι χώρες BICS μπορούν να αποτελέσουν τη λύση αλλά μπορούν να αποτελέσουν και πρόβλημα. Γιατί αν η οικονομική μηχανή αρχίζει ε, και σκοντάφτη, όπως ενδεχομένως θα αρχίσει να συμβαίνει στην Ινδία και την Κίνα τα επόμενα χρόνια. Ε, αυτό θα επηρεάσει ε, πολιτικά και στρατιωτικά όλη την περιοχή. Για παράδειγμα, ανάμεσα ε, στην Κίνα και την εθνικιστική της, τον εθνικιστικό παροξισμό και στους γειτόνους της υπάρχουν εντάσεις. Ορισμένες χώρες της ΑΣΕΑΝ, ε, η Ιαπωνία και η Ινδία για παράδειγμα, συμμαχούν για να εξορροπήσουν την ισχύ της Κίνας. Ε, μια σύγκρουση στην περιοχή της, ε, του Ειρηνικού και της Ασίας θα αποτελούσε πρόβλημα για όλο τον κόσμο. Στον Ατλαντικό ωκεανό δεν έχουμε τέτοιου είδους συστημικές απειλές. Ε, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών ανάμεσα στην Νότιο Αμερική, την Αφρική και την Ευρώπη ε, ε, όμως δεν θα μπορούσε να καταπολεμηθεί χωρίς τη συμμετοχή της Βραζιλίας. Η Βραζιλία επίσης θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια, στην τροφιμική ασφάλεια και στις κλιματικές αλλαγές τα επόμενα χρόνια. Οπότε αυτές οι χώρες, οι BRICS πλήν της Ρωσίας, δεν είναι οι ηγεμονικές χώρες του αύριο. Καμία από αυτές δεν πουλάει ένα εναλλακτικό παγκόσμιο όραμα, ε, ούτε ε, αυτή τη στιγμή καμία από αυτές επιθυμεί ε, να επικρατήσει τον κόσμο. Τώρα, σε 50 χρόνια δεν ξέρω τι θα γίνεται. Θέλουν όμως να έχουν φωνή στις μεγάλες αποφάσεις που παίρνονται στον κόσμο και επιθυμούν οι κανόνες του παιχνιδιού να προσαρμοστούν στα συμφέροντά τους. Θα τελειώσω λέγοντας ότι αυτές οι αναδυόμενες χώρες γνωρίζουν πολύ καλά πως αν ο, όποιος δεν είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι στο μενού που τρώνε. Ε, οπότε οι παραδοσιακές ε, δυνάμεις ε, θα πρέπει να το δεχτούν ε, αλλά να υπενθυμίσουν κιόλα σε χώρε BRICS ότι όποιο είναι στο τραπέζι πρέπει να πλένει και τα πιάτα μετά και να μαγειρεύει κιόλα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ακούσουμε τον Άντριου Σμόλ στη συνέχεια. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η ακρόαση αυτή αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη σε σχέση με τις επιπτώσεις των αναδυόμενων δυνάμεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπε και ο συνάδελφος, δεν μπορούμε να μιλάμε για μια ενιαία πολιτική έναντι των ε, BRICS, αλλά θα πρέπει να, βρούμε, να δούμε τους ευρύτερους στόχους και τα διασταυρούμενα στοιχεία για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να έχουμε κάποια γνώση σε σχέση με αυτές τις πολιτικές που δεν είναι αλληλένδετες ως προς την Κίνα, Βραζιλία, Ρωσία και ούτω καθεξής. Θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ε, ρόλο σε αυτή τη μεταβατική πορεία και δεν θα πρέπει να υποβαθμιστεί ο ρόλος της. Εάν όμως τα επόμενα χρόνια ε, δεν λάβουμε θέση, τότε θα μας βάλουν στην άκρη. Επίσης, θα πρέπει να δούμε τα, την κλινορομιά τη, της ε, μη ε, ευθυγράμμισης με μία συγκεκριμένη πολιτική γενικότερα, αλλά η Κίνα διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο και αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Τέλος, ίσως μιλάμε για μια στρατηγική χωρών ρυθμιστών ή χωρών που διαδραματίζουν ένα καταλητικό ρόλο. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι χώρες οι οποίες πραγματικά επηρεάζουν τα τεκτενόμενα και οι αποφάσεις τους έχουν επιπτώσεις ανά τον κόσμο. Κατά πόσο λοιπόν μπορούμε να μιλήσουμε για ένα πολυμερές σύστημα το οποίο ε, δεν άπτεται άμεσα με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη είναι στην εμπροστοφυλακή αυτής της μεταβατικής θέσης. Στο άνω μέρος της κορυφής βρίσκονται οι ΙΠΑ και η Ευρώπη όμως μπορεί με το όραμά της ως προς την παγκόσμια τάξη πραγμάτων να προβάλλει συγκεκριμένες θέσεις και προκλήσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βρούμε μια στρατηγική εξισορρόπηση με βάση τις νέες αυτές δυνάμεις. Τη στιγμή όμως που όλα εξαρτώνται από ένα αλληλένδετο παγκόσμιο σύστημα ως προς τις μεταφορές, την προσφορά, τη ζήτηση, τις προμήθειες και την σταθερότητα των περιοχών, η Ευρώπη αναλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο έργο, είτε μέσω αρρωγής στρατιωτικών δυνάμεων, χρηματοδοτήσεων, πολυμερών οργανώσεων και ούτω καθεξής. Και δεν ξέρουμε κατά πόσο θα επιταχύνουν το βήμα οι αναδιόμενες χώρες. Όμως, εξαιτία του ειδικού βάρους της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προβάλλει συγκεκριμένα στοιχεία. Όπως ξέρουμε, Ω ε, ως προς τη μεταφορά τεχνολογίας, η, Ινδία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, όμως η Κίνα δεν μπορεί να έχει το ίδιο. Αυτό θα είχε στρατηγικές συνέπειες. Η πλεονεκτική μας θέση είναι ότι διαδραματίζουμε σημαντικό ρόλο παγκοσμίω. Δηλαδή, ποιος θα κάθεται στο τραπέζι στο μέλλον. Όλα αυτά τα στοιχεία η τεχνολογία, οι δυνάμεις στην παγκόσμια σκακέρα και ούτω καθεξής διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Αυτό που μας ενδιέφερε δυστυχώς περισσότερο ήταν να ασκήσουμε δύναμη και όχι η θέση που κατέχουμε και πώς μπορούμε να επηρεάσουμε τα πράγματα. Δηλαδή ε, μέσα στους G20 είδαμε δυστυχώς ότι ο ρόλος μας δεν ήταν καταλυτικός. Δυστυχώς μπορούν να αλλάξουν αυτά τα πράγματα, αλλά αυτή η ευκαιρία συρρυκνούται και δυστυχώς θα παραμεριστούμε εάν δεν δράσουμε. Δεύτερον, οι χώρες BRICS, όπως είπε και ο συνάδελφος, είναι μία αποκλεινόμενη ομάδα. Δηλαδή δεν είναι μία ομοιογενής ομάδα. Υπάρχουν ε, πέρα από τις ΗΠΑ, η Ιαπωνία, ε, Κορέα, Ιαπωνία και BRICS, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε να κάνουμε με τις 20 μεγαλύτερες οικονομίες μαζί με την Τουρκία. Η Ρωσία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά, όπως είπε και ο συνάδελφος. Όμως οι άλλες έχουν κοινά στοιχεία και η Κίνα και Ινδία και η Βραζιλία θα θεωρηθούν υποανάπτυξη χώρες αν και αποκτούν ειδικό βάρος. Το περιορισμένο τους ΑΕΠ θα είναι αρκετά χαμηλό και στο μέλλον. Άρα θα πρέπει να καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες έτσι ώστε να μην αναλάβουν μεγάλα φορτία διεθνώς τη στιγμή που αντιμετωπίζουν εσωτερικές δυσχέρειες αυτό το στοιχείο ε, σχετίζεται με μια πολιτική um, μια πολιτική που σχετιζόταν με τον μπλοκ των αδεσμεύτων. Γι' αυτό πιστεύω ότι μέσα στα πλαίσια της ε, ολοκλήρωσης θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι και πώς θα έχει αυτή η μετάβαση γιατί υπάρχουν χώρες που δεν θέλουν να είναι ουραγοί της δύση μέσα στα πλαίσια των οικονομικών ε, συμφερόντων της δύση και δεν θέλουν να ολισθήσουν προς αυτή την κατάσταση. Το είδαμε με την ε, Λιβύη, ε, με την Βυρμανία και ούτω καθεξής. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι κατά πόσο μπορεί να γίνει μία διαχρονική διευθέτηση. Δηλαδή υπάρχουν ξεχωριστά συμφέροντα των αναδιόμενων χωρών, όμως υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία μέσα στα πλαίσια των πολυμερών σχέσεων. Η Κίνα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Υπάρχει αμοιβαία κατανόηση, υπάρχουν κοινά συμφέροντα, αλλά δεν υπάρχει σύγκληση ως προς τις κοινέ αξίες, την ε, δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα ή τον ολοκληρωτισμό. Επειδή έχει ειδικό οικονομικό και πολιτικό βάρος η Κίνα, αποτελεί μια ξεχωριστή κατηγορία για μας. Δεν σημαίνει ότι δεν θα προβεί σε επιλαγές που θα συμβαδίζουν με τις δικές μας, αλλά όπως ισχύει με το Ιράν, Σουδάν και Λιβύη, όλα αυτά θα γίνουν μετά από υπολογισμό και μία συνένεση η οποία δεν θα αφορά μόνο τη Δύση. Πώς μπορούμε να καλύψουμε, δηλαδή πώς μπορούμε να φτάσουμε σε αυτή τη ε, συνένεση ως προς αυτές τις χώρες ρυθμιστές. Ως προς την Ινδονησία, Ινδία, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούν αυτές οι χώρες να μεταβούν προς το δικό μας πεδίο, το δικό μας στρατόπεδο. Όμως υπάρχουν στρατηγικές επιλογές. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο θα κινηθούν προς μία κατεύθυνση μέσα στα πλαίσια της πολυμέρειας και κατά πόσο αυτό θα έχει επιπτώσει στο διεθνές σύστημα. Τώρα, ως προς τη μόχλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να λάβουμε σαφείς αποφάσεις για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις επιλογές. Θα πρέπει να μπορέσουμε να δούμε ποιες χώρες θα είναι υποστηρικτές του συστήματος ως προς την επέκτασή τους στον οικονομικό, ε, πολιτικό τομέα, τομέα άμυνας, τεχνολογιών και ούτω καθεξής. Και να δούμε κατά πόσο μπορούμε να προωθήσουμε τα στρατηγικά τους συμφέροντα. Κατά πόσο μπορούμε να συνεργαστούμε με τη νέα γενναία αρχηγών και κυβερνήσεων. Ίσως να μην έχουμε ε, βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, αλλά ο καρπός αυτών των ε, προτεραιοτήτων και στοιχείων θα φανεί. Δυστυχώς πολλές αυτές οι χώρες θα μπορέσουμε τι χώρε αυτές θα τι ε, επηρεάσουμε μέσω μόχλευσης. Ως προς τη Ρωσία και την ε, Κίνα θα πρέπει να δούμε πώς θα κινηθούμε καθώς και με την ε, Ινδία, Βραζιλία και Ινδονησία για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε και τις επιλογές της Κίνας. Εάν δεχτούμε αυτή την προσέγγιση θα ενισχύσουμε τις θέσεις μας με τις ΗΠΑ και την Κίνα. Πολύ περισσότερο. Το ζήτημα είναι κατά πόσο είμαστε μέσα στο στρατηγικό παιχνίδι. Η Κίνα δέχεται αυτή τη σοβαρότητα, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι κατά πόσο μπορούμε εμείς να δράσουμε στα ε, παγκόσμια πεπραγμένα επηρεάζοντάς τα θα πρέπει να προβάλλουμε μία στρατηγική για αυτές τις χώρες ρυθμιστές για να δούμε κατά πόσο αυτές οι χώρες θα συγκλίνουν προς τις δικές μας αξίες και συμφέροντα. Bene, apriamo il primo giro di domande. Γύρος ε, ερωτήσεων. Πέτερλε. Κύριε Πέτερλε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, οφείλω να ομολογήσω ότι ανησυχώ περισσότερο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό τον καιρό και λιγότερο για τις χώρες BRIC. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχώ. Άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά αυτά που είπατε για τη στρατηγική μας και πώς ε, την εξηγήσατε, τη στρατηγική που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι σε αυτές τις χώρες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω Σύμφωνα με τις αναλύσεις σας, έχετε διαπιστώσει καμία αλλαγή σε ό,τι αφορά την έννοια και την αντίληψη των χωρών αυτών για την εξουσία. Θέλουν να έχουν το μερίδιο τους στην εξουσία ή ήδη από τώρα βλέπουν το ειδικό τους βάρος κάπως διαφορετικά και πώς βλέπετε τη συνεργασία με τις χώρες αυτές. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Νομίζω ότι και οι δύο ομιλητές θα μπορούσαν ενδεχομένως να μου απαντήσουν. Ξεκίνησαν από τη ε, υπόθεση ότι αυτές οι νέες ενδυνάμει ομάδες ε, δεν θα αντιμετωπίσουν ε, μεγάλα προβλήματα. Βεβαίως η Κίνα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μεγάλα οικονομικά προβλήματα λόγω του υψηλού χρέους της. Αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μια γραμμική πορεία και για, για όλες αυτές τις χώρες της ομάδας. Εάν λοιπόν ξεκινήσουμε από την υπόθεσή σας αυτή, οι αναδυόμενες αυτές δυνάμεις θα αποτελέσουν πηγή ανασφάλειας για τις υγιές Άρα μιλάμε για μια πολιτική εξισορρόπησης ε, ε, δυνάμεων μέσα στα πλαίσια ε, παπιλούμενου καταστάσεων. Θεωρείτε ότι ελοχεύει ένας τέτοιος κίνδυνος, δηλαδή έστω και, έστω και κατά να προκύψουν αυτές οι ενδεχόμενες σειράξεις. Όσον αφορά τη Ρωσία, από πλευράς ε, Δυτικής Ευρώπης αλλά και Κεντρικής, η Ρωσία αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα διότι προσπαθεί να ορίσει τους κανόνες και να τους επιβάλλει και στις ε, γείτονες χώρες, κάτι το οποίο μας φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση. Έχουν το λόγο... Α, με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος. Ο κύριος Άτκινς έχει το λόγο. Πρόεδρε, σε σχέση με τα όσα είπε ο συνάδελφος Σόπφριν και συνεχίζω από εκεί, κάτι που δεν ρωτήσαμε ακόμα είναι το εξής. Αν γίνει μια σύγκριση με τις Ηνωμένε Πολιτείε που υποτίθεται ότι έχει μια ε, στάση απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο, με την έννοια ότι αν υπάρχει κάποια σύγκρουση ε, συμμετέχουν για να ε, αποτρέψουν κάποια σύραξη ή διαφορά. Αλλά πώς θα βλέπατε εσείς την ε, Κίνα ή την Ινδία ή και άλλους στο προσεχές μέλλον θα μπουν σε αυτό το παιχνίδι ή μήπω είναι ήδη εκεί. Οι απαντήσεις λοιπόν από τους δύο μιλητές. Ποιος θα ήθελε το λόγο πρώτος. Θα προσπαθήσω να απαντήσω την ερώτηση αυτή. Ως προς τα προβλήματα της Κίνας, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν νομίζω ότι η κινέζικη οικονομία είναι βιώσιμη, διότι εξαρτάται από τον υπόλοιπο κόσμο και την καλή υγεία του υπόλοιπου κόσμου και δεν νομίζω ότι ε, βοηθάμε ιδιαίτερα γιατί είμαστε αλληλένδετοι. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Οι ίδιοι οι Κινέζοι λένε ότι για να υπάρχει μια βιώσιμη οικονομία θα πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη εγχώρια αγορά στην ίδια την Κίνα. Αυτό σημαίνει όμως ένα μεγάλο και ισχυρό δίκτυο κοινωνικής πρόνοιας που σημαίνει ότι θα βγουν πολλά χρήματα από το δίκτυο επενδύσεων να καταπολεμηθεί η διαφθορά και ούτω καθεξής. Και σημαίνει απελευθέρωση πιστώσεων. Εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο, μάλλον ε, αν γίνει κάτι τέτοιο, σταματά λίγη το κομμουνιστικό καθεστώς στην ε, Κίνα. Δεν μπορούμε να χαρούμε βεβαίως γι' αυτό, γιατί αν πέσει η Κίνα θα πέσουμε και όλοι οι υπόλοιποι, διότι είμαστε αλληλένδετα εξαρτώμενοι. Δεν είναι δηλαδή πρόβλημα μόνο δικό μας, θα είναι πρόβλημα, μάλλον δεν θα είναι πρόβλημα μόνο της Κίνας, αλλά θα είναι και δικό μας και τον είπα και ούτω καθεξής. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να ε, λυθεί συλλογικά. Τώρα, Εάν υπάρχει πρόβλημα στην Κίνα, τότε θα υπάρξουν δυνατότητες επέκτασης ενδεχόμενων σειράξεων αν ξεκινήσουν από εκεί. Δεν ισχύει το ίδιο με τη Βραζιλία, διότι στη Βραζιλία δεν υπάρχει συστημικός κίνδυνος προβλημάτων ασφαλείας. Η Ρωσία αποτελεί πρόβλημα Το ζήτημα είναι πώς μπορούν να συμβαδίσουν η Ρωσία, η Κίνα, η Βραζιλία και η Ινδία. Αλλά η ε, Ρωσία δεν εντάσσεται εδώ. Βρίσκεται κάπου αλλού. Δεν συμβαδίζει με την Κίνα, την Ινδία και τη Βραζιλία. Ως προς την ανταγωνιστικότητα και τη συνεργασία. Ο κύριος Πέτερλε ε, υπέβαλε αυτό το ερώτημα, δηλαδή κατά πόσο συνεργάζονται και πόσο ανταγωνίζονται. Εξαρτάται από το αντικείμενο. Υπάρχει υψηλός ανταγωνισμός, ε, μιλώ για τη Βραζιλία, διότι η βιομηχανία της Βραζιλίας ανησυχεί με τις εισαγωγές προϊόντων από την Κίνα. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός η Ινδία δεν είναι ανταγωνιστής της Βραζίλιας. Εξαρτάται λοιπόν για ποια χώρα μιλάμε και για ποιο προϊόν, για ποια αγαθά. Υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας ή ανταγωνισμού. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω και να δούμε ποιος ανταγωνίζεται ποιον. Όταν η Apple και η Nike πουλά προϊόντα τα οποία συναρμολογούνται στην Κίνα, τότε ποιος ανταγωνίζεται την Ευρώπη, η Apple ή η Κίνα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σίγουροι, να δούμε δηλαδή πώς λειτουργούν οι βιομηχανικές αλυσίδες, ποιος κάνει τη συναρμολόγηση, ποιος παίρνει τα χρήματα. Όλοι ξέρουμε το iPod συναρμολογείται, φτιάχνεται στην Κίνα και οι Κινέζοι παίρνουν 10% της προστιθέμενης αξίας και η Apple 60%. Άρα ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο κακός. Πολλές εξαγωγές της Κίνας στην Ευρώπη γίνονται από μεγάλες πολυεθνικές που πουλούν στην Ευρώπη και πολλά προϊόντα που εξάγουμε συναρμολογούνται αλλού. Άρα θα πρέπει να μιλήσουμε για την γεωγραφία της παραγωγής. Γιατί θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να μιλούμε πια για ανταγωνισμό χώρων. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, είναι πεθαμένο αυτό το σχήμα. Έχει λήξει. Μιλάμε για πολυεθνικές που επεκτείνονται παντού. Θα πρέπει να γίνει μια μεγάλη μελέτη για το πώς λειτουργεί αυτή η οικονομία. Είναι μια αλληλένδετη οικονομία. Ο κύριος ε, Πασκάλ Λαμή στον ΠΟΕ έχει κάνει μια μεγάλη εκστρατεία επί του θέματος. Λέει ότι θα πρέπει να επανακαταρτήσουμε τις στατιστικές γιατί δεν ξέρουμε ποιος κερδίζει και ποιος χάνει σε αυτόν τον αλληλένδετο κόσμο. Να σχολιάσω μερικά πράγματα κι εγώ. Καταρχήν σε ό,τι αφορά τη γραμμικότητα. Ναι, είναι αλήθεια θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο κάποια από αυτές τις ε, χώρες ε, να δουν την οικονομία τους να αλλάζει πορεία. Ε, είναι και αυτές ευαίσθητες, αλλά δεν πρέπει να κάνουμε και το αντίστροφο λάθος. Έχουμε προβλέψει εδώ και, προβλέπουμε εδώ και πολύ καιρό την κατάρρευση της Κίνας λόγω χρέους, πλην όμως αυτό έχουμε διαψευστεί. Ε, ενδεχομένως θα συμβεί το γεγονός αυτό της κατάρρευσης τα επόμενα 20-30 χρόνια αλλά μπορεί η ανάπτυξη της ε, Κίνας να συνεχιστεί στα ίδια επίπεδα για πολύ καιρό. Τώρα σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο πολέμου. Ακόμα και σήμερα υπάρχει το θέμα. Στην θάλασσα της Νότιας Κίνας, για παράδειγμα, υπάρχει ο κίνδυνος. Τις τελευταίες δύο μέρες μιλούσα για την περίπτωση περιορισμένου πολέμου μεταξύ Κίνας και Βιετνάμ ε, εξαιτίας ε, ενδεχομένως ε, κάποιου λάθους ή λανθασμένου υπολογισμού. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και θα πρέπει να τον δεχτούμε ως κάτι υπαρκτό στο μέλλον. Το ίδιο θα απαντούσα και για το θέμα της Ρωσίας. Η Ρωσία είναι σε διαφορετική κατηγορία από μόνη της. Ακόμα και όταν ε, μιλάμε για χώρες που αποτελούν ρυθμιστικό παράγοντα, ε, η, ο ρόλος της Ρωσίας είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Ε, η αποτελεσματικότητά μας ε, στο χειρισμό της Ρωσίας διπλωματικά είναι πολύ διαφορετικό πράγμα από ότι ο διπλωματικός χειρισμός της Κίνας. Ε, σε ό,τι αφορά την, τον ηγεμονικό ρόλο αυτό των κρατών στο μέλλον, ε, αν θα είναι εμπεριαλιστικά κράτη ή όχι. δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή Έχουμε δει διαφ... αλλαγέ στη στάση ό,τι αφορά τι αρχέ, για παράδειγμα, τη μη επέμβαση. Ε, η Κίνα θα γίνει στρατιωτική ισχύ, στρατιωτικά ισχυρή χώρα και θα προστατεύει τα συμφέροντά τη, έστω και εκτό ε, ακόμα και εκτός της επικράτειάς της, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει υπεριαλιστική δύναμη. η σημερινή της ε, στάση εξαρτάται από μια σχετική αδυναμία που είχε στο παρελθόν. Ε, δεν νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει. Η Κίνα, για παράδειγμα, στην ε, Λιβύη έχει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να δράσει ούτε στρατιωτικά, ενδεχομένως ούτε και διπλωματικά. Αυτό νομίζω δεν θα ισχύσει στο μέλλον. Ε, δεν θα ισχύει στο μέλλον και η Ινδία θα γίνει στρατιωτική δύναμη η οποία θα μπορεί ε, να αναλαμβάνει επιχειρήσει σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Τώρα, αν έχει αλλάξει η ισορροπία δυνάμεων. Ε, νομίζω ότι ναι, έχει γίνει αλλαγή στην ισορροπία δυνάμεων, ιδιαίτερα μετά την οικονομική κρίση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την Κίνα Νομίζω ότι ε, έχουμε βρει μια καινούργια ισορροπία ε, στον, στο αντιληπτό βάρος της κάθε χώρας και ε, η, ήδη η, αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ποια θα είναι η ισχύ σε αυτών των χωρών τα επόμενα δέκα χρόνια. Οπότε στο μυαλό μας αρχίζουμε και προβλέπουμε και ε, προεξοφλούμε τις αλλαγές που θα γίνουν στην ισορροπία των ε, ισχύω τα επόμενα χρόνια. Ε, τουλάχιστον αν δεν αλλάξει η δυναμική των πραγμάτων. Σε αυτή την περίπτωση η ε, η ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωση θα επηρεαστεί και αυτή και ενδεχομένω πιο νωρίς και από την οικονομία. Ε, Οι κύριοι Ναν και η Στισοάια ζήτησαν να λάβουν το λόγο επί του θέματος. Ο κύριος Τάνοκ ζήτησε το λόγο. Καταρχήν θέλετε τώρα να παρέμβετε ή θέλετε να ακούσετε τους, του, τους ε, άλλους εισηγητές για να ακούσετε και να ίσως ενδεχομένως να υποβάλλετε την ερώτησή σας μετά. Σύριλ Ναν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω γερμανικά. Επιτρέψτε μου να προσθέσω μερικά στοιχεία από τη σκοπιά ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις σχέσεις με τις χώρες BRICS αλλά και την κάθε μία χώρα ξεχωριστά από τις χώρες BRICS. Πρώτον, το εμπόριο με τις χώρες BRICS για μια χώρα σαν τη Γερμανία ε, ε, έχει πολύ μεγάλη σημασία και εκρήγνεται. 30% ας πούμε αυξάνεται το εμπόριο με την Κίνα, με την Ινδία, με τη Βραζιλία. 15% ε, του παγκοσμίου εμπορίου πλέον είναι αυτές οι χώρες και στο μεταξύ 18% του γερμανικού εξωτερικού εμπορίου Προπενταετία ήταν το μισό, 8 με 9%. Διπλασιάστηκε λοιπόν το εμπόριό μας με τις χώρες αυτές. Αυτές οι χώρες έχουν όλες μια κοινή ε, θέση, ε, ένα συμφέρον, ε, ερευνητική, οικονομική συνεργασία, ακαδημιακή συνεργασία, πανεπιστημιακή. Σε άλλου αυτό είναι πιο έντονο, όπω είναι η Κίνα, αυτό εκφράζει έντονα. Άλλοι είναι λίγο πιο επιφυλακτικοί, πάντω είναι κοινό για όλε τι χώρε. Όλες αυτές οι χώρες είναι σημαντικοί μας σύμμαχοι στη Γερμανία και συνομιλητές για θέματα όπως ε, είναι θέματα αλλαγής κλίματος ή ολοκλήρωση του γύρου της ε, Ντόχα. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια τώρα για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης κρατών BRICS από τη σκοπιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενός κράτους μέλους. Με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι μεμονωμένες χώρες όπως η Γερμανία έχουν κάνει στρατηγικές εταιρικέ σχέσεις και διεξάγουν στρατηγικό διάλογο. Μια χώρα όπως είναι η Κίνα έχει 15% των συναλλαγματικών της αποθεμάτων σε ευρώ. Αυτό είναι καλή είδηση. Επίσης, κάνουμε και διαπραγματεύσουμε την Ινδία για μια ζώνη ελευθέρων συναλλαγών. Ταυτόχρονα όμως διαπιστώνουμε ότι η Ευρώπη δεν είναι καλά προετοιμασμένη για τις σχέσεις της με τις χώρες αυτές. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλές εταιρικέ σχέσεις, στρατηγικές σχέσεις με πολλές χώρες του κόσμου. Ε, καλύτερο λοιπόν να έχουμε λιγότερες για να είναι περισσότερο το αποτέλεσμα. Less is more. Δηλαδή ας επικεντρωθούμε σε αυτές τις χώρες που είναι πολύ σημαντικές, να μην έχουμε με όλους στρατηγικές σχέσεις. Στη συνέχεια, υπάρχει μεγάλη διαφορά ε, στη στάση ε, μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών. Η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ δραστήρια, ενώ η ΕΙΕΔ ε, ε, το ε, Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περισσότερο τρικλοποδιές βάζουν ένα στον άλλον παρά έχουν αποτέλεσμα. Δεν είναι αυτό ούτε ικανοποιητικό ούτε ευπρόσδεκτο για τη Γερμανία και προσπαθούμε να κάνουμε προτάσεις αλλά και αυτές γνωρίζουν τα όρια τους. Σε αυτό το πεδίο σίγουρα θα χρειαστεί δράση. Οι χώρες BRICS κοιτούν και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τις διμερείς μας σχέσεις και θεωρούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα δυνητικά σημαντικό εταίρο, αλλά έναν εταίρο που προς το παρόν είναι η δεύτερη επιλογή τους. Προηγείται η διμερής σχέση με τα κράτη. Γιατί δεν οργανώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως θα θέλαν οι χώρες BRICS και από πλευράς οικονομίας, επενδύσεων, ε, έρευνας, ε, δεν μιλάει με την ίδια φωνή θα πρέπει να το προωθούμε και ως Γερμανία εμεί πάντα ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτό. Πού βρίσκεται η Ευρώπη, γιατί απουσιάζει, γιατί δεν είναι ακόμα εδώ που την περιμένουμε και θα έπρεπε να είναι. Και ένα τρίτο που θα ήθελα σύντομα να αναφέρω είναι η στάση των χωρών BRICS στα Ηνωμένα Έθνη. Γνωρίζετε ότι αυτό το καιρό ε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας γίνεται ε, συμμετέχουν ε, ε, η Νιγηρία, όλες οι χώρες BRICS και ε, τέσσερις από το Συμβούλιο και ο Ινδός πρέσβης είπε ότι επίκυνται αλλαγές και η Ινδία σε δύο χρόνια δεν θα αποχωρήσει από το Συμβούλιο Ασφαλείας, θα θέλει να διατηρήσει την έδρα της. Βέβαια, η κατάσταση είναι κάπως διαφορετική. Οι χώρες BRICS στα Ηνωμένα Έθνη υποστηρίζουν η μία την άλλη. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συμμαχία Βραζιλίας, Ινδίας για παράδειγμα. Αυτό όμως είναι αντίβαρο απέναντι στη Δύση ή μήπως είναι αμυντική στάση τους αυτή η συμμαχία η απάντηση δεν είναι τελείως μονοσήμαντη ούτε ξεκάθαρη. Αυτό που είναι σίγουρο ότι στη Νέα Υόρκη σιγά σιγά βλέπουμε να συνασπίζονται οι χώρες BRICS σε επιμέρου θέματα. Το είδαμε και για τη Λιβύη αλλά και για τη Σύρια που ουσιαστικά δεν έχουν ε, ενδιαφέρον ε, ε, οι χώρες BRICS να βγει ψήφισμα από το Συμβούλιο ασφαλεία και επίση η Ινδία στα Ηνωμένα Έθνη ε, τη συνεργασία και τη σχέση της με την Κίνα για να κερδίσει και τη εμπιστοσύνη της. Γιατί ξέρουμε ότι η Κίνα είναι από τις πέντε χώρες που έχουν ε, ε, δικαίωμα βέτο και γίνονται συζητήσεις να διευρυνθεί αυτό. Επίσης, η ΙΠΣΑ που είναι η Ινδία, Βραζιλία και η Αφρική επίσης συνεργάζονται πιο στενά και θέλουν να ε, ενισχύσουν το ειδικό βάρος ε, των BRICS και ε, σε σχέση με ένα εξάμεινο πριν, η Αμερικανική κυβέρνηση είπε ότι θα ενδιαφερόταν πολύ για το ψήφισμα της Συρίας να συμμετέχουν και χώρες BRICS και να συμμετέχουν ενώντας να συμπαραταχθούν με τη Δύση στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτή είναι νέη τόνη, νέο ύφο. Μέχρι τώρα δεν χρησιμοποιεί το, τέτοιο ύφο στα Ηνωμένα Έθνη. Εν πάση περιπτώσει, στα Ηνωμένα Έθνη και πάλι είναι διχασμένοι, είναι ε, ε, από τους, πέντε BRICS, οι δύο είναι μόνιμα μέλη στο Συμβούλιο Ασφαλείας, οι άλλοι τρεις όχι. Ε, ακόμα δεν έχει λυθεί το θέμα των μονίμων μελών, βεβαίως ξέρετε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Τι είναι. Ο κύριος Τάνοκ έχει το λόγο για να υποβάλει ερώτηση. Τίποτα δεν με πείθει ότι οι χώρες BRICS έχουν να κάνουν με ε, εσωτερική συνοχή. Αποτελούν ένα μεγάλο οικονομικό μπλοκ, μάλλον ένα συμπίλημα χωρών που θα μπορούσαν να είναι ε, μεγάλοι παίκτες, αλλά ε, ειδικά η Κίνα και η Ινδία είναι μεγάλοι εχθροί. Ο κύριος Σμολ μου υπενθύμησε ότι ίσως δεν θα πρέπει να άρουμε το εμπάργο προς την Κίνα επί του παρόντος. Το θέμα αυτό είχε συζητηθεί στο Κοινοβούλιο εδώ και δέκα χρόνια και τότε είχαμε συμφωνήσει. Η ε, Ρωσία έχει να αντιμετωπίσει μια μεγάλη δημογραφική κρίση, κάτι το οποίο θα έχει επιπτώσεις από οικονομικής και στρατιωτικής πλευράς ε, μακροχρόνια. Κάτι που είναι εντελώς αντίθετο με την κατάσταση της Κίνας, Ινδίας και Ινδονησίας. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ή ορισμένα κράτη-μέλη όπως και το Ηνωμένο Βασίλειο ε, χορηγούν βοήθεια προς την Ινδία και την Κίνα. Θα πρέπει να δίνουμε τη βοήθεια ανάλογα με το συνολικό ΑΕΠ και όχι το κατακεφαλή. Πολλοί συνάδελφοι, ιδιαίτερα στην ε, Επιτροπή, uh, στην Επιτροπή της ε, ΑΦΕΤ, όπου θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη συνοχή, πιστεύουμε ότι σε έναν κόσμο πολλαπλών πόλων θα μπορούσαμε να ε, δράσουμε έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια πιο δυνατή ένωση. Αυτό μπορεί να ισχύει και για τις χώρες BRICS και η Βραζιλία θεωρεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, πραγματικό ε, στη διεθνή ε, σκακέρα ή θεωρείτε ότι σε 10 χρόνια θα έχει εξαφανιστεί. Ε, τώρα αυτό που μας απασχολεί βεβαίως το άμεσο μέλλον είναι η Ευρωζώνη και η επιβίωσή της. Το λόγο έχει ο κύριος Μόρα Μπεναβέντε. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Χαίρομαι που είμαι εδώ προσκλήθηκα να σας παρουσιάσω μια διαφορετική οπτική γωνία, την οπτική γωνία ενός κράτους μέλους σε σχέση με την ομάδα των χωρών BRICS. Πριν πω στο θέμα μου, θα ήθελα να κάνω δύο διευκρινιστικά σχόλια. Πρώτον, θα αναφερθώ στις χώρες BRICS με ένα πιο ευρύ τρόπο. Θα περιλάβω και χώρες όπως το Μεξικό ή Νότιος Αφρική. Καμία χώρα που αποτελεί περιφερειακή ε, δύναμη ε, υπ' αυτή την έννοια. Για ποιο λόγο το κάνω αυτό. Θα το δείτε αφού ολοκληρώσω την παρουσίασή μου, θα το καταλάβατε, ελπίζω. Δεύτερο σχόλιο. Θα σας παρουσιάσω την ισπανική οπτική γωνία βέβαια, αλλά σύμφωνα με τις συζητήσεις που έχουμε συναδέλφους στην Ευρώπη και αλλού, ε, ε, έχω την εντύπωση ότι αυτή η άποψη συμπίπτει με την άποψη πολλών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέραν της Ισπανίας. Λοιπόν, διμερείς συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις χώρες BRICS. Αυτή η σχέση αποτελεί σημαντικό κομμάτι ε, της εξωτερικής πολιτικής οποιοδήποτε κράτου μέλους. Θα πρέπει να κάνουμε την εξής υπόθεση εργασίας. Η εξωτερική πολιτική του κάθε κράτους μέλους ε, θα αλλάξει με την θέση ισχύ της συνθήκης Λισαβόνας ανεξάρτητα των επιθυμιών του κράτους μέλους, ανεξάρτητα της πολιτικής βούλησης του κάθε κράτους μέλους. Έχουμε μπει σε, μια καινούργια, ε, σε ένα καινούργιο θεσμικό σε μια καινούργια θεσμική πραγματικότητα ε, και θα αλλάξει. Τώρα πώς θα αλλάξει θα το δούμε αργότερα. Ε, έχουμε μια καινούργια θεσμική δομή λοιπόν, η οποία θα επηρεάσει τις εξωτερικές πολιτικές των κρατών μελών. Τώρα, με ποιον τρόπο. Η απάντηση είναι η εξή, πολύ απλή. Με τον τρόπο που θα χρειαστεί έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει ένας αξιόπιστος, ε, σεβαστός παίκτη στην παγκόσμια σκαγέρα. Οι χώρες BRICS αντιλαμβάνονται τις διεθνείς σχέσεις ως σχέσεις ισχύω και επιρροής. Ε, θα πρέπει λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι αξιόπιστος παίκτη, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να κάνει τίποτα στις σχέσεις με τις χώρες BRICS. Συνεπώ, δεδομένου ότι χρειάζονται λοιπόν να αλλάξουν οι εθνικές εξωτερικές πολιτικές ε, τι απομένει στη σχέση ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις χώρες BRICS. Οι χώρες BRICS είναι χώρες ε, σημαντικές στις, ειδημερείς σχέσεις με, τη, με χώρες όπως η Κίνα ή η Βραζιλία ε, περιλαμβάνουν ε, μια ευρία γκάμα θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, στρατηγική σχέση, πολιτική σχέση, οικονομική σχέση όλο και περισσότερο, ένα τεράστιο δυναμικό στον πολιτιστικό τομέα κλπ. Με τέτοιες χώρες, με τέτοια μεγέθη χωρών, η εξωτερική πολιτική λοιπόν περιλαμβάνει μια σειρά τομέων. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας, με την ανάγκη αλλαγών των εθνικών εξωτερικών πολιτικών, ε, θα πρέπει να συμβιβαστούμε σε επίπεδο κρατών μελών. Να δούμε ε, τα διάφορα θέματα τα οποία έθιξα στις στρατηγικές σχέσεις για παράδειγμα. Αυτές οι χώρες, Κίνα, Βραζιλία, Μεξικό, είναι χώρες κλειδιά για να λύσουμε, ή για να αντιμετωπίσουμε, να χειριστούμε οποιοδήποτε πρόβλημα που επηρεάζει την παγκόσμια κοινότητα. Είτε πρόκειται για την ε, κλιματική αλλαγή, τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, το, την μεταρρύθμιση του διεθνούς νομισματικού ε, συστήματος, χρηματοπιστωτικού συστήματος κλπ. Χωρίς αυτές τις χώρες δεν μπορεί καν να ξεκινήσει μια συζήτηση για αυτά τα παγκόσμια προβλήματα. Σε τέτοιου είδους λοιπόν ζητήματα τα, η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των θεσμικών της οργάνων πρέπει να είναι ο μοναδικός συνομιλητής εξ όλων μας, γιατί δεν, δεν έχει πλέον κανένα νόημα ε, μεμονωμένα το κάθε κράτος ε, μέλος να ακολουθεί μια εθνική πολιτική για τέτοιου είδους ζητήματα στατική σημασία. Ε, είτε σε διμερεί σχέσει είτε στα, στα πολυμερή φόρα. Κάτι τέτοιο θα αποδυνάμωνε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης της θέσει τη Ευρωπαϊκή αλλά θα ήταν και μη ρεαλιστικό. Συνεπώ, κατά την άποψή μου, όλα αυτά τα στατική σημασία θέματα είναι θέματα τα οποία άπτονται τις δράσεις τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο ισχύει και για τις περιφερειακές συγκρούσεις. Και εδώ είναι λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα. Μέση Ανατολή, Ναγκρόνο Καραβάχ, Σάχελ, Σομαλία. Και εδώ ο μόνος δυνατός συνομιλητής με τις χώρες BRICS είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των θεσμικών της οργάνων. Και εδώ έχουμε δύο διαφορετικά, δύο διαφορετικά ζητήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δράσει ως διαμεσολαβητής και αυτό είναι ένας σημαντικός πολιτικός ρόλος που μπορεί να παίξει. Και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να αναλάβει αυτό το ρόλο. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παγκόσμιο στερέωμα. Οπότε αναμφίβολα θα πρέπει να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά υπάρχει κι άλλο ένα ζήτημα σχετικό με τις περιφερειακές συγκρούσεις. Ε, οι επεμβάσεις, στρατιωτικές ε, επεμβάσεις, ε, οι οποίες απαιτούν χρήση ε, στρατιωτικού προσωπικού, ακόμα και πολιτών, εμπειρογνωμόνων κλπ. Και πάλι αυτή η παρουσία μπορεί να ενισχύσει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, περνάω στις πολιτικές σχέσεις, διμερείς πολιτικές σχέσεις. Εδώ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Και εδώ μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο είδου σύγκρουση ανάμεσα στα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Η δική μου άποψη είναι σαφή. Τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, έχουν ε, αξιόλογε και ουσιαστικές μόνιμες διμερείς σχέσει με τις χώρες BRICS. Για πολλούς λόγους. Ένας λόγο είναι η ασφάλεια. Ε, με την συνθήκη της ε, Λισαβόνας κάναμε ένα ουσιαστικό βήμα μπρος στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Αλλά ε, η, ε, κανένας δεν μπορεί να πει ότι όλες, όλα τα προβλήματα ασφάλειας των κρατών μελών καλύπτονται από την συνθήκη της Λισαβόνας. Όχι, ούτε και αυτός ήταν ο στόχος. Συνεπώς, αν κάτι πάει στραβά και ένα κράτος μέλος βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση, μπορεί να αναμένει ελεγγύη από τα κρατη αλλά τίποτα από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, αλλά τίποτα παραπάνω. Συνεπώ, οποιοδήποτε μυρογνωμόνο θα σα έλεγε ότι σε τέτοιου περιπτώσει είναι σημαντικό η κάθε χώρα να διαθέτει ουσιαστικέ μερεί σχέσει με τι μεγάλε πρωτεύουσε. Για παράδειγμα, το Πεκίνο. Αυτό που χρειαζόμαστε όμως είναι διαφάνεια, σαφήνεια, ε, αλλά οι διμερείς σχέσεις πρέπει να είναι ουσιαστικές με τις χώρες BRICS. Με την επιφύλαξη βέβαια του ρόλου που θα δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα θεσμικά της όργανα. Τώρα, τρία συμπεράσματα για την έκθεσή σας. Πρώτον, η συνθήκη Λισαβόνας επιφέρει, θα έπρεπε να επιφέρει σημαντική αλλαγή στην εθνική εξωτερική πολιτική των κρατών μελών. Αυτός θα είναι βασικός κανόνας του παιχνιδιού στο μέλλον. Δεύτερον, με τις χώρες BRICS η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ο μοναδικό συνομιλητής σε ζητήματα παγκόσμιας εμβέλεια. Και βέβαια αυτά περιλαμβάνουν την παγκόσμια διακυβέρνηση. Τρίτον, τα κράτη-μέλη θα διατηρήσουν και ενδεχομένως θα εμβαθύνουν κιόλα τις διμερείς του σχέσεις με τις χώρες BRICS. Αλλά αυτές οι διμερείς σχέσεις θα πρέπει να είναι διαφανείς, να εξασφαλίζεται πλήρη διαφα... πλήρης διαφάνεια και σεβασμό στο ρόλο των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Bene, l'ultimo intervento. παρέμβαση είναι του κυρίου Βιορέλ Ιστιτσοάια. Ε, κάθε φορά ε, δυσκολεύουν πάρα πολύ να προφέρω σωστά τα ονόματα. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που τουλάχιστον προσπαθείτε να προφέρετε το όνομά μου. Ακόμα και οι συμπατριώτες μου αντιμετωπίζουν τη Θα προσπαθήσω και εγώ να συνεισφέρω σε αυτή τη συζήτηση του πάνελ ενώπιον της ΑΦΕΤ. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και επειδή είμαι ο τελευταίος ε, που λαμβάνει το λόγο, έχω το ευεργέτημα να έχω ακούσει τι ε, προείπαν οι άλλοι και σε ποια σημεία στάθηκαν. Επειδή όμως εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, θα πρέπει να πω ότι ε, είμαι πολύ υπερήφανος διότι θα πρέπει να καλύψω θέματα που σχετίζονται με τους τέσσερις ε, στρατηγικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ιδιαίτερα την Κίνα και την Ινδία και ε, ως προς την δημοκρατία της ε, Κορέας και την Ιαπωνία δεν εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Όπως ξέρετε, οι χώρες BRICS είναι μια πολύ χαλαρή ομάδα και αυτό μέσα στα γενικότερα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Οι χώρες είχαν να αντιμετωπίσουν πολλές ε, προκλήσεις, γι' αυτό θεώρησαν ότι αυτή η ομαδοποίηση θα ήταν κάτι το πολύ θετικό για να έχουν μεγαλύτερη ισχύ διεθνώς. Γιατί μιλάμε για πόρους, ε, δύναμη, μέγεθος και ούτω καθεξής. Επειδή θα σας μιλήσω για τον προγραμματισμό μας, και πώς θα δράσουμε από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να αναγνωρίσω ότι διαχωρίζονται σε διάφορα γεωγραφικά σχήματα και ομαδοποίησεις ανάλογα με τις γεωγραφικές συνθήκες και τις περιστάσεις. Έχουμε κοινή προσέγγιση μεν, υπάρχει κάτι το κοινό, δηλαδή αυτός ο τίτλος που ε, δόθη εδώ και μερικά χρόνια για λόγους αυρότητας ίσως. Οι συνάδελφοι στο πάνελ έθιξαν πολλά και σημαντικά ζητήματα, αλλά νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με διαφορετικά σχήματα και τμήματα που ασχολούνται με αυτό τον προγραμματισμό. Θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι ήδη από πέρυσι υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για να ορίσουμε το περιεχόμενο αυτής της στρατηγικής εταιρικής σχέσης. μέσα στα πλαίσια της κατάρτισης της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πολύ σας τα ε, είπατε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ασχολήθηκε ε, με τρεις στρατηγικούς εταίρους, δηλαδή την Κίνα, τη Ρωσία και την Ινδία. Και ε, μελλοντικά θα ασχοληθούμε και με την Ινδία και τη Βραζιλία που βρίσκονται σε αυτή την άτυπη ομάδα. Πρόκειται για μία άτυπη ομαδοποίηση όπως και όπως σας είπα ήδη. Δεν πρόκειται για επιλογή αυτών των χωρών. Ομαδοποιήθηκαν για συγκεκριμένους λόγους. Γιατί η διεθνής συγκυρία κατέδειξε ότι ίσως θα είχαν να ωφεληθούν εάν ομαδοποιούντο μέσα στα πλαίσια της αμοιβαίας υποστήριξης. Πρόκειται για αναδιόμενες δυνάμεις, περιφερειακές ή διεθνείς και ίσως να έχουν πολλά να μάθουν ή μεν από τις δε, να αναφερθούν στις εμπειρίες τους, στους διεθνείς οργανισμούς και θεωρώ ότι βρίσκονται σε μία καμπή Μπορεί βεβαίως να μετατραπούν και μετατρέπονται βαθμία σε μεγάλους οικονομικούς παίκτες. Πρόκειται για μια διαδικασία μαθητείας. Είναι ένα κληροδότημα του παρελθόντος και επειδή στο παρελθόν ασχοληθήκαμε διμερώς με αυτές τις χώρες, είδαμε ότι φτάσαμε σε μία ατζέντα διμερών σχέσεων, ένα οικοδόμημα διμερών σχέσεων με συγκεκριμένα μέσο και μακροχρόνια προγράμματα και μηχανισμούς διαλόγου. Πρόκειται για ε, μία συγκεκριμένα σχήμα χαλαρής στρατηγικής, χαλαρών στρατηγικών. Δεν νομίζω όμως ότι μπορούμε να τις ομαδοποιήσουμε και να τις ε, αντιμετωπίσουμε σαν ένα ενιαίο μπλοκ. Όσοι μελετήσουν περισσότερο τις, σχέσεις, τις οικονομικές σχέσεις και εμπορικές σχέσεις στους ε, διεθνείς οργανισμούς και φόρα, μπορούν να διαπιστώσουν και συγκρούμενα συμφέροντα, εάν λάβουμε υπόψη περιφερειακά ή εθνικά συμφέροντα. Κληρονομήσαμε λοιπόν και θα κρατήσουμε για λίγο αυτή τη βασική ατζέντα όπως έχει συγκροτηθεί και τους μηχανισμούς για πολιτικό διάλογο, διασκέψεις ε, κορυφής σε τακτά χρονικά διαστήματα ως προς τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον πρόεδρο του Συμβουλίου, ο οποίος ε, μπορεί να εκπροσωπήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο υψηλότερο επίπεδο για να αποστείλει συγκεκριμένα μηνύματα. Η πρώτη επίσκεψη του Προέδρου του Συμβουλίου κατά τα μέσα Μαΐου στην ε, Κίνα απέδωσε καρπούς. Είδαμε ότι η Κίνα μπορεί να συνεργαστεί κατά νέο τρόπο να ορίσουμε νέες προτεραιότητες ανάλογα και με τα ενδιαφέροντα των κρατών μελών αλλά και σε συλλογικό επίπεδο. Μπορούσαμε λοιπόν να ορίσουμε νέες προτεραιότητες και ένα νέο πεδίο συνεργασίας μέσα στα πλαίσια της ετήσιας διάσκεψης που θα γίνει αργότερα φέτος. Θα ήθελα να πω ότι η ίδια η υπηρεσία μέσα στα πλαίσια του διαλόγου σε τακτά χρονικά διαστήματα εξερεύνησε τις οδούς που είχαν διανοιχθεί στο παρελθόν μέσω του δικτύου διμερών σχέσεων, ε, δηλαδή ε, συνεργασία οικονομικής εταιρικής σχέσης, όπως είχε οριστεί στο παρελθόν, είχαμε αρκετά καλά αποτελέσματα και με την ε, Δημοκρατία της Κορέας με βάση την εμπορική συμφωνία η οποία συνήφθη φέτος τον Ιούλιο και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε και μια πολύ ε, καλή ε, εμπορική συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με την Ινδία. Επίσης μπορούν να συναυθούν και πολιτικές συμφωνίες μέσα στα πλαίσια των εταιρικών οικονομικών σχέσεων. Κατά τα μέσα Ιουνίου είχαμε ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων με την Κίνα, καθώς και άλλες συζητήσεις όπως τον διάλογο σε τακτά χρονικά διαστήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι μιλάμε για πάγιες αξίες και γιατί ορισμένες χώρες εκπλήσονται από το πώς αντιμετωπίζουμε τη δική τους τοπική πραγματικότητα. Επειδή λοιπόν ασχολούμαστε με αυτές τις χώρες από πλευράς στρατηγικών εταιρικών σχέσεων, και όπως προείπαν οι συνάδελφοι, ίσως εγώ θα πρέπει να το δω από λίγο διαφορετική οπτική γωνία. Νομίζω ότι υπάρχουν συγκεκριμένα εκτενή ε, στοιχεία με βάση τις ε, διμερείς σχέσεις καθώς και τις ε, στρατηγικές εταιρικές σχέσεις. Ίσως μπορούμε να κινηθούμε πέραν των διμερών σχέσεων και να διερευνήσουμε ενδεχομένως και τις σχέσεις αυτές και τους συσχετισμούς για να δούμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις προσδοκίες στο δικό μου τουλάχιστον τμήμα, δηλαδή ως προς την Ασία, Κίνα και Ινδία, ίσως φτάσουμε σε πολύ καλές εταιρικέ σχέσεις, απλώς θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ε, για το ποιο θα είναι το σημείο εκκίνησης. Βεβαίως η, ε, η Κίνα είναι μια ευρύτατη οντότητα και ίσως θα πρέπει να το δούμε το θέμα υπό πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες. Επίσης είναι εντελώς διαφορετική η κατάσταση στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική, στην Χερσόνησο της Νότιο-Ανατολικής ε, Ασίας και ούτω καθεξής. Είδαμε πώς ε, ε, απομακρύνθηκαν και οι πολίτες, οι πολίτες μας από τη Λιβύη και αυτό δείχνει ότι μπορούν να δράσουν και οι τοπικοί φορείς μέσα στα πλαίσια αυτών των δυνατοτήτων. Ως προς τις περιφερειακές πολιτικές, είπαμε ότι ορισμένες περιφέρειες έχουν ένα ειδικό βάρος και επειδή είναι σημαντική στρατηγική εταίρη και επειδή θέλουμε οι εταίροι αυτοί να εξακολουθήσουν να είναι σημαντικοί, μας ενδιαφέρει πώς θα προωθήσουμε τις πολιτικές μας σε αυτές τις περιφέρειες. Ο Πίτερ Μάντελσον είχε πει μερικά χρόνια ότι μπορούμε να διαμορφώσουμε το μέλλον ανάλογα με το πώς θα μεταχειριστούμε την Κίνα. Δηλαδή πώς μπορούμε να προωθήσουμε μία σχέση με αυτό τον βασικό παγκόσμιο παίκτη. Μας ενδιαφέρουν οι μακροχρόνιες εταιρικές σχέσεις. Αυτό θα πρέπει να το διερευνήσουμε. Άκουσα πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις από εσάς και γι' αυτό ήθελα και εγώ να συμμετάσχω και προγενέστερα στις απαντήσεις. Θα ήθελα να σας πω ότι πέρσι ε, λέχθη ότι, χρειάζ, ότι υπάρχουν εταιρικές στρατηγικές σχέσεις, αλλά τώρα χρειάζεται μια γενικότερη εταιρικότητα. Χαίρομαι για τη συζήτηση εδώ στην ΑΦΕΤ. Ελπίζω να μπορέσω και εγώ να αντλήσω από τη δική σας σοφία. Ο κύριος Κέλλαμ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους σας. Ήταν συναρπαστική η συζήτηση και πάρα πολύ μεγάλη ανταμοιβή για όλους μας έτσι. Η βασική έννοια εδώ είναι η αυξημένη αλληλεξάρτηση. Κανείς δεν μπορεί να την αποφύγει. Ούτε το επιθυμεί. Η απάντηση θα είναι όμως ενισχυμένη συνεργασία και ε, συντονισμός. Έχει γίνει αντιληπτό το μήνυμα, οι χώρες BRIC θέλουν να έχουν μεγαλύτερο λόγο ε, και μεγαλύτερο βάρος και βαρύτητα στην παγκόσμια οικονομία και στην παγκόσμια πολιτική. Το θέμα όμως είναι πώς θα γίνει αυτό. Ακριβώς επειδή χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία και μεγαλύτερο συντονισμός, αυτό μπορεί να γίνει μόνο, ας πούμε, αυξάνοντας το κράτος δικαίου στη διεθνή πολιτική. Τι σημαίνει αυτό. Μεγαλύτερη διαφάνεια, ίσες ευκαιρίες, αμοιβαιότητα, όσο και μείωση της διαφθοράς. Άλλος τρόπος να γίνει αυτό είναι να προσπαθεί κανείς να αυξήσει το στρατιωτικό και πολιτικό ρόλο κάθε αναδυόμενης δύναμης. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια σαφής ε, διαφωνία, ε, διαίρεση μάλλον από τη μια έχουμε την Κίνα και τη Ρωσία που αυτό προσπαθούν να κάνουν και από την άλλη την Ινδία και τη Βραζιλία που δεν το πράττουν. Και σε ό,τι αφορά την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επανειλημμένα ο κύριος Σμόλ μίλησε για την ευκαιρία που είναι ε, προσωρινή και θα κλείσει αυτό το παράθυρο της ευκαιρίας όπως λέγεται. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν επίσης το θέμα είναι ε, αν θα αντιδράσει συντονισμένα ή αν θα εκμεταλλευτεί ή θα αξιοποιήσει διμερείς σχέσεις που έχει με κάθε χώρα μπρήξε χωριστά. Και νομίζω ότι ο Ισπανικός συνάδελφος πρότεινε μια πάρα πολύ καλή φόρμουλα ότι οι διμερείς σχέσεις θα πρέπει να είναι πολύ πιο διαφανείς αλλιώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να διαδραματίσει τον παγκόσμιο ρόλο της ή να αυξήσει την αξιοπιστία της. Έρχομαι τώρα στο ερώτημά μου. Υπάρχει όμως ε, αρκετή πολιτική ενθάρρυνση και οικονομική παρότριση και κίνητρα για να συνεργάζονται περισσότερο και να ανταποκρίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο συντονισμένα. Συμφωνώ ότι ε, πρέπει να βγάλουμε τη Ρωσία. Είναι big, δεν είναι brick. Γιατί η Ρωσία είναι πραγματικά ιδιάζουσα περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ. Μη μου... Ο συνάδελφος Βαν παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω του ομιλητέ. Ακούσαμε και αποκλήσει απόψεων και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Uh, ε, μπερδεύτηκα λίγο από αυτά που είπε ο κύριος Μπενεβέντε. I'm not quite sure what you were saying. Ε, δεν κατάλαβα πολύ καλά τι λέτε, διότι από τη μια μας λένε συνέχεια ότι το περιεχόμενο της ΚΕΠΑ είναι αυτό που της προσδίδουν τα κράτη-μέλη. Δηλαδή δεν έχει αυτόνομη ζωή ό,τι επιθυμούν και προερούνται τα κράτη-μέλη να θεωρήσουν κοινή εξωτερική πολιτική είναι η ΚΕΠΑ. Από την άλλη μας λέτε όμως ότι μετά τη σύνθηκη της Λισαβόνας και τη θέση σε ισχύ που κατά τα άλλα ε, παρόδο δεν έχει δημοκρατική νομιμοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας μην τρέφουμε αυτά πάτες. Ε, λέτε ότι το κράτη μέλη τώρα είναι υποχρεωμένα να αλλάζουν την εξωτερική τους πολιτική λόγω ε, εξαιτία τη συνθήκη Λισαβόνα. Δηλαδή τώρα ε, είναι μια κοινή μας υποχρέωση. Δεν ξέρω, αυτά τα δύο στοιχεία είναι μάλλον αντιφατικά μεταξύ τους. Θα μπορούσατε λίγο να μας διευκρινίσετε um, τη θέση σας. Η Γερμανία, ας πούμε, τι θα θεωρούσε αν της λέγατε να σταματήσει τις διμερείς σχέσεις πολύ ε, αμφιβάλλω κατά πώς θα ευδοκιμήσει. Επίσης φαίνεται να δείχνεται μεγάλο ε, ενθουσιασμό ε, για την ΕΠΑ. Μα οι επιχειρήσεις στη Λιβύη έδειξαν πόσο φρούδα και κενή είναι αυτή η πολιτική, έως και ανύπαρκτη. Αυτό που προσπαθούμε είναι να θέλουμε να βρίσκουμε μια εξωτερική πολιτική και πολιτική αμήνης και μετά να προσαρμόζουμε την πραγματικότητα ε, σε αυτό το γκορσέ για να ανταποκρίνεται στις δικές μας επιθυμίες και αυτά που λέμε. Για παράδειγμα στην ΕΠΑΑ η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε ε, να κάνει τα Ηνωμένα Έθνη να συμφωνήσουν με κάποιο είδου ανθρωπιστική αποστολή στη Λιβύη, απεγνωσμένα μάλιστα, ε, και να εντάσσεται αυτό στην ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Ουδή το ήθελε αυτό. Μετά απεγνωσμένα προσπάθησε να προχωρήσει σε ναυτικό αποκλεισμό. Και αυτό δεν το ήθελε κανεί. Αφήσαμε λοιπόν τα Ηνωμένα Έθνη και πιάσαμε το ΝΑΤΟ. Γιατί, διότι το πρόβλημα είναι ότι μόνο τα μισά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ συνεισφέρουν στην αποστολή γιατί συνεχώς ε, ε, υπάρχουν διάφορες άλλες ε, καταστάσεις που τους αποσπούν την προσοχή και ασχολούνται με αυτές. Λοιπόν, σε σχέση με τα όσα συζητούμε σήμερα, ποια είναι η σχέση μεταξύ της εμπορικής πολιτικής και της εξωτερικής πολιτικής. Ιστορικά, και είναι ενδιαφέρον αυτό, τα κράτη συχνά κατάφεραν να τα κρατήσουν χωριστά. Αν κοιτάξετε πώς οδηγηθήκαμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Βρετανία αγόραζε από τη Γερμανία χημικά για παραγωγή πυρομαχικών. Ακόμα και μετά την έναρξη του πολέμου, νομίζω, για κάποιο διάστημα συνέχισε. Δηλαδή, άλλο εμπορική πολιτική, άλλο η εξωτερική. Και υπάρχουν πολλά άλλα ιστορικά παραδείγματα. Σας ερωτώ λοιπόν σήμερα, ποια είναι η σχέση εμπορικής με την εξωτερική πολιτική. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Βανόρντεν. Ο κύριος ε, Ξύπ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ένας από τους τελευταίους ομιλητές, ο κύριος Μπουντούρα, ο τελευταίος ομιλητής μας ε, έκανε μια πολύ καλή σύνοψη μίλησε για στρατηγικές εταιρικές σχέσεις ε, με χώρες του ομίλου BRICS. Θα πρέπει όμως τώρα να δούμε ποια θα είναι η στρατηγική μας, ποια στρατηγική θα εκπονήσουμε. Και αυτή η δήλωση δείχνει ότι εμείς ήμασταν οι οπισθοφυλακοί σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζονται αυτές οι αναδυόμενες χώρες και οι χώρες που γνωρίζουν πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Δεν ξέρουμε ποια είναι τα στοιχεία διασύνδεσης. Ακούσαμε ότι η Ρωσία δεν θα έπρεπε καν να ανήκει σε αυτή την ομάδα. Και ίσως, ίσως θα έπρεπε, ίσως όχι να ενταχθεί. Όλες οι χώρες γνωρίζουν πολύ καλά τις ικανότητές τους, τη δύναμή τους και προσπαθούν να κάνουν και επίδειξη δύναμης. Ανταγωνίζονται δε και σε αυτόν τον τομέα και αυτό το βλέπουμε σε διάφορους τομείς. Θυμάμαι μία συνομιλία που είχαμε έναν Πολωνό πρέσβη στην Κίνα κατά τα τέλη της δεκαετίας του 80 τότε ρώτησε έναν πρωθυπουργό από την Ανατολική Ευρώπη πώς βλέπετε να εξελίσσεται η χώρα σας κατά την επόμενη εκατονταετία. Και η απάντηση ήταν «Μα δεν προγραμματίζουμε τόσο μακριά». Δεν έχουμε τόσο μακροχρόνιο προγραμματισμό. Νομίζω ότι πολλά αποκαλύπτει αυτή η απάντηση. Δείχνει και την πολιτική όπως καταρτίζεται από τις κινέζικες αρχές. Δεν έχουν τόσο μακρόπνοα σχέδια. Αυτό το ζήτημα το συζητήσαμε και εδώ αλλά και σε άλλες επιτροπές, ιδιαίτερα ως προς το θέμα της ασφάλειας της ε, προμήθειας ε, πρώτων υλών. Βλέπετε ότι το 80 με 90% ε, των, των, πηγών βρίσκονται στην Κίνα ως προς τις σπάνιες γιές. Επίσης, η Κίνα έχει και άλλα αποθέματα, όπως τον ενεργειακό τομέα. Αυτό αφορά βεβαίως και τη Ρωσία. Και βλέπετε ότι και στη Βραζιλία τα αποθέματα ενέργειας αναπτύσσονται με ταχύ ρυθμό και ίσως αλλάξει κατάσταση άρδιν στο εγγύς μέλλον και να είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου η Βραζιλία. Βεβαίως ίσως το δημογραφικό είναι ένα από τα κοινά στοιχεία με τη Ρωσία. Τα πράγματα βεβαίως δεν είναι και τόσο καλά ως προς το ρωσικό μέτωπο, όμως πρόσφατα άκουσα ότι θα επέλθουν μεγάλες δημογραφικές αλλαγές σε όλες αυτές τις χώρες τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή η Ινδία θα προτρέξει της ε, Κίνας ως προς την γεννητικότητα και αυτό αφορά και την ε, Νιγηρία. Βεβαίως και εκεί υπάρχει θέμα ενεργειακών, ενεργειακών προμηθειών και γι' αυτό ίσως αλλάξει και το παιχνίδι συσχετισμών στην Αφρική. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τι γνώμη έχετε για το ποιος θα κατέχει αρχηγική θέση σε αυτό το πακέτο στο μέλλον. Ίσως αλλάξει η δυναμική και ο συσχετισμός δυνάμεων στην ομάδα όπως προανέφερα και ίσως καιροφυλακτούν και μεγάλες κρίσεις. Ποιος λοιπόν θα κατέχει αρχηγική θέση στην ομάδα αυτή στο μέλλον. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι η, στρατηγικές, η στρατηγική εταιρική σχέση με αυτές τις χώρες καθώς και οι εμπορικές συμφωνίες. Είδαμε ότι ως προς τις εμπορικές ε, συμφωνίες υπάρχει μεγάλο εμπορικό έλλειμμα με άλλους εταίρους, όπου, όπως το Μερκοσούρ, όπου υπάρχει μεγάλο εμπορικό έλλειμμα. Και τώρα μιλώντας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αρχές, αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι τι επιπτώσεις θα υπάρχουν ως προς τις σχέσεις μας με αυτές τις χώρες. Ο κύριος Λαντσμπέργκης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ένα μόνο σχόλιο. Αν θα είναι BRIC ή big. Ε, ως ε, νέοι παγκόσμιοι ε, πρωταγωνιστές. Και συχνά αποκαλούνται αναδυόμενες οικονομίες αυτές παγκοσμίω. Αλλά το να τις αντιμετωπίζουμε μόνο ως αναδυόμενες οικονομίες δεν είναι αρκετό. Δηλαδή δεν είναι σωστό, δεν είναι το μόνο κοινό τους χαρακτηριστικό. Βεβαίως Εάν κύριος και θεός μας είναι η οικονομία, ε, όπως έλεγε ο Καρ Μάρξ, τότε εντάξει, ναι, είναι αξιοσημείωτο, αλλά υπάρχουν και άλλα στοιχεία που μετρούν τη σημασία ενός κράτους. Όπως είπε και ο συνάδελφος Ξύπ, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και θα ήθελα να τις δω αυτές τις χώρες και να σε εκτιμήσω ως αναδυόμενες δημοκρατίες και όχι οικονομίες μόνο. Και δύο είναι μεγάλες αναδυόμενες δημοκρατίες. Πάντα τονίζουμε ότι η Ινδία είναι τόσο σημαντική δημοκρατία. Επίσης, δεν θα, θε... θα θέλαμε να τις δούμε όλες τις χώρες αυτές να μπαίνουν στο δημοκρατικό κόσμο και να τον ενισχύουν με την παρουσία τους. Αυτή η γραμμή είναι πάρα πολύ σημαντική για το μέλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τη διατηρήσουμε αυτή τη γραμμή και να μην σβηστεί από οποιαδήποτε δουαλιστική ε, αντιμετώπιση, να κάνουμε το BRICS αυτό ένα μίξ και να δούμε τι θα βγει. Όχι. Να έχουμε κάποιους ε, γνώμονες στη δουλειά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, με τη σειρά Ναν Μπεναβέντε και Μπουντούρα για να απαντήσουν. Ευχαριστώ. Ως προς το ερώτημα του κυρίου Βανόρτεν, είναι ένα θέμα που μας απασχόλησε στη γερμανική κυβέρνηση. Μας απασχολεί συχνά ποιες είναι οι σχέσεις εμπορικής, εμπορικών πολιτικών και πολιτικής εξωτερικών σχέσεων. Τι γίνεται όταν υπάρχουν πλεονάσματα με ορισμένες χώρες και πώς μπορούμε να αρχίσουμε μια συζήτηση που δεν επιθυμούν. Και αυτό άπτεται του θέματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από την ε, εμπειρία μας βλέπουμε ότι αυτοί οι, μάλλον οι οικονομικές σχέσεις πρέπει να διέπονται από ένα υγιές πλαίσιο, αλλά βεβαίως υπάρχει και ο συσχετισμός με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ιδιαίτερα οι Κινέζοι φίλοι μας ακούν πολύ προσεκτικά όταν διακυβεύονται τα δικά τους συμφέροντα. Έχουν μεγάλο συμφέρον στην μεταφορά τεχνολογιών, στις επενδύσεις. Εκεί θέλουν να μάθουν τα πάντα από την Ευρώπη για να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τότε υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα για να ακούσουν ζητήματα που δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Δέχονται υποδείξεις από την κυρία ε, Μέρκελ τη στιγμή που ε, απευθύνεται στον Πρωθυπουργό της Κίνας κατά ένα συγκεκριμένο τρόπο ενώπιον δημοσιογράφων. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ποια είναι τα, τα συμφέροντα των μεν και των δε και μετά υπάρχει αυτή η διάδραση. Έχουμε να μάθουμε και εμείς πολλά για να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση γιατί διαφορετικά υπάρχουν δύο μονόλογοι και ούτε καν. Τώρα, επανερχόμενος στα ανθρώπινα δικαιώματα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και οπωσδήποτε στη δική μας, αυτό είναι το επίκεντρο των μελημάτων μας. Θέλουμε λοιπόν να ε, δώσουμε αυτή τη μάχη σε καθημερινή βάση κατά επιτυχή τρόπο ή δυνατόν, τη στιγμή που έχουμε επιχειρήματα υπέρ ημών. Αυτές είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα των σχέσεων μας με την Κίνα και το ίδιο ισχύει και για την ε, Ινδία και με την Ινδία. Ως προς το ερώτημα του κυρίου Κέλαμ, θα ήθελα να πω ότι οι χώρες BRICS έχουν ε, υψηλά κίνητρα για αυτή τη διάδραση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Και θεωρούμε ότι αυτή η διάδραση είναι κάτι που θα προτιμούσαν χώρες όπως η Κίνα από τις χώρες BRICS. Αλλά αυτό είναι δυνατόν είναι όταν υπάρχει ένας πραγματικός εταίρος. Υπάρχει. Ε, λοιπόν, υπάρχουν αυτά τα αμοιβαία συμφέροντα και γι' αυτό υπάρχει και αυτός ο διάλογος με την Κίνα. Και με την Ινδία αντιμετωπίζουμε, έχουμε την ίδια ακριβώς, τα ίδια ακριβώς δεδομένα. Ευχαριστώ. Το πρώτο τμήμα της ερώτησης του κ. Φανόρδεν ε, αφορά το εξή. Εγώ θα πω την άποψή μου με λίγο διαφορετικό τρόπο. Με τη συνθήκη της Λισαβόνα δεν αλλάξαμε τον τρόπο διαμόρφωσης των πολιτικών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωση. Δεν αλλάξαμε τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνουμε την εξωτερική μας πολιτική. Αυτό που άλλαξε είναι το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο παρουσιάζεται αυτή η πολιτική στον υπόλοιπο κόσμο και μέσα στο οποίο διαχειριζόμαστε αυτή την πολιτική. Ε, η λογική πίσω από αυτό δεν νομίζω ότι είναι ε, που δεν είναι ομοσπονδιακή λογική. Η λογική είναι ότι ο κόσμος μας γίνεται όλο και πιο πολυπολικός. Οπότε είναι καλύτερο ε, να έχουμε μία ενιαία φωνή. Είναι καλύτερο να εκπροσωπούμαστε από έναν άνθρωπο. Οπότε αυτό που λέω είναι ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προσαρμόσουν τις εθνικές πολιτικές προς αυτήν την κατεύθυνση. Αν η συνθήκη της Αβώνας δίνει, αναθέτει την πλήρη εκπροσώπηση μια συγκεκριμένη κοινή εξωτερικής πολιτικής σε έναν ή δύο συγκεκριμένη περίπτωση άτομα και ταυτόχρονα δημιουργούμε μια καινούρια δομή την υπηρεσία εξωτερικών δράσεων, εξωτερική δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα πρέπει και κάθε χώρα να προσαρμόσει τη δική τη εξωτερική πολιτική. Γιατί αλλιώ τα κράτη-μέλη θα πάψουν να, είναι, να έχουν ισχυρό λόγο. Ε, αν, αν ε, ε, κάποιος είναι μέλος τη Συμβουλίου Ασφαλεία, θα πρέπει να έχει θέση για όλα τα ζητήματα ε, της παγκόσμιας, ε, τα, πολυγιώτα παγκόσμια ζητήματα. Όμως αυτό δεν ισχύει για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Η δική μου εμπειρία είναι ότι όλοι περιμένουν να δουν πώς θα λειτουργήσει ο θεσμός του υπατού εκπροσώπου και της επίσης εξωτερικής δράσης. Ε, για μας όλα αυτά είναι κάτι δεδομένο, δεδομένο, αλλά για τον υπόλοιπο κόσμο δεν είναι. Περιμένουν, ε, κρατούν μια ε, επιφυλακτική στάση προς το παρόν. Ε, η ανάγνωση όμως της συνθήκης αβώνας μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τις εξωτερικές πολιτικές. Γιατί δεν είναι δυνατόν να διατηρείται εθνική πολιτική πέραν της πολιτικής που εκφράζεται στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να καταλήξουν σε μια ενιαία στάση. Σε αντίθετη περίπτωση θα υποσκάπταμε ακριβώς όλο αυτό το οικοδόμημα το οποίο έχουμε φτιάξει. Ε, ε, Ευχαριστώ. Ειλικρινά πιστεύω ότι οι ερωτήσεις σας ε, πραγματικά αντανακλούν μια πάρα πολύ μεγάλη κατανόηση της κατάστασης που αντιμετωπίζουμε από πολλές πλευρές. Είπαμε ότι χωρίς χώρες BRICS εμφανίζονται να πρωταγωνιστούν αισθητά και σε περιφερειακό επίπεδο και σε παγκόσμιο. Και θα πρέπει να αλλάξουμε και εμείς την ατζέντα μας, να καλωσορίσουμε ε, τις φιλοδοξίες τους με την καλή έννοια πάντα και να τονώσουμε και τη συμμετοχή τους γιατί έχουν πολλούς πόρους και χώριους πόρους για να μπορέσουν να διαμορφώσουν ε, και νέες καταστάσεις και νέα καθεστώτα διεθνώς. Ορισμένοι παρατηρητές είδαν την Κίνα να είναι κάπως συγκρατημένος επιφυλακτικός διεθνός ε, εταίρος. Πάντως τα τελευταία χρόνια, ε, τις δύο τελευταίες δεκαετίες και μετά και την επιτυχία των Ολυμπιακών Αγώνων το 2008 του Πεκίνου, πήρα μια γεύση του τι σημαίνει να έχεις μια νέα ε, στάση και συμπεριφορά στα παγκόσμια τεκτενόμενα και στη διαμόρφωση των διαφόρων διεθνών οργανισμών. Βεβαίως εσείς γνωρίζετε καλύτερα από μένα τα προβλήματα ε, που απορρέουν από την ε, οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, πόσο έφεραν στην επιφάνεια την Κίνα και πόσο η ίδια δέχτηκε πολλές προκλήσεις και διεθνείς ε, προσδοκίες και έχει ταυτόχρονα και πολλά ζητήματα να αντιμετωπίσει όμω και εσωτερικά και εξωτερικά, όπω και το θέμα τη συναλλαγματική ισοτιμία. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, θα έλεγα ότι για εμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη, σε πολλέ περιπτώσει. Και τώρα έχουμε και στο G20 μια νέα συνεργασία. Έχουμε πεδίο ακριβώ να δράσουμε, να πιέσουμε, να χρησιμοποιήσουμε κάποιου μοχλούς βέβαια Εσεί θα κρίνετε αν στο G20 η Ευρωπαϊκή Ένωση υποεκπροσωπείται ή υπερεκπροσωπείται ή έχει τη σωστή εκπροσώψη. Σε ό,τι αφορά τη δική μα υπηρεσία, ε, πρέπει να σα πω ότι θεωρούμε ένα πολύ καλό βήμα το G20 να συνεργαζόμαστε με τι χώρε αυτέ. Και σε περιφερειακό επίπεδο υπάρχουν πολλά ζητήματα από τα οποία μπορούμε να επωφεληθούμε αν συνεργαζόμαστε σωστά με τι χώρε αυτέ. και σωστά τονίστηκε ότι έχουν πολλού πόρου που επηρεάζουν όχι μόνο τις ε, διεθνείς και περιφερειακές αγορές, αλλά και κάποιες αλυσίδες ε, προμήθειας ε, υλών και κάποιο κόστος. Αν αύριο κάποιες από τις χώρες αυτές, αλλά κυρίως η Κίνα, ανακοινώσει ότι διπλασιάζει, τριπλασιάζει τις εισαγωγές κάποιου αγαθού, αυτό θα διαταράξει σοβαρά τις διεθνείς αγορές και ο τρόπος με τον οποίο ε, εμείς ε, καταλαμβάνουμε κάποιες θέσεις και τοποθετούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση διεθνώς θα είναι προς όφελος και της Ένωσης και των κρατομελών και του κόσμου. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα τέλος πιστεύω πάρα πολύ ότι είναι σημαντική εταίρη ε, αυτή διεθνώς και θα πρέπει λίγο να ανακυκλώσουμε θα έλεγα, για να να αναδιατυπώσουμε τελείως τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για να είναι πιο αποτελεσματική. Δηλαδή, να θέτουμε υπόψη τους τα συμφέροντά μας και το ενδιαφέρον μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις χώρες αυτές. Όπως πολύ σωστά είπε κάποιος συνάδελφος του πάνελ, πολλά πράγματα διακυβεύονται εκεί. Και συχνά Καταρχήν, ε, αυτοί οι εταίροι θέλουν ίση μεταχείριση. Δεν θέλουν ε, ανταντάγματα. Ε, και όχι μόνο, αν δεν είναι ίση με εμά, πολλέ φορέ θέλουν να αναγνωρίζονται ω πρωταγωνιστέ. Δεν θα πρέπει να πηγαίνουν να του κάνουμε κήρυγμα όπως γινόταν πριν από δεκαετίες υπό όρου μέχρι και πρόσφατα, δεν νομίζω ότι θα έχει αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα όμως όπως είπε και κάποιος στο νέο πλαίσιο μετά τη Λισαβόνα, για τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε ένα νέο πλαίσιο, μπορούμε να διαβιβάζουμε τα μηνύματά μας με άλλο τρόπο σε πολλούς αποδέκτες με πολλά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας γιατί οι κοινωνίες με τον τρόπο που λειτουργούν έχουν πολλούς διάβλους για να αλληλεπιδρούμε με αυτούς τους εταίρους είτε είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις, πανεπιστήμια, ακαδημίες. Πολλά φόρα, πολλά μέσα, πολλά κανάλια που βοηθούν τις κοινωνίες να εξελίσσονται και να ασπάζονται και τις δικές μας αξίες. Σας ευχαριστώ. Allora, l'ultima replica è del relatore Valladao. Θα ήθελα και να, να, στην ερώτηση του κύριου Τάνοκ σε σχέση με τις σχέσεις Βραζιλίας-Ευρώπης και το καθεξής. Ως προς την βοήθεια προς την Ινδία, Κίνα, Βραζιλία, αυτό αποτελεί ένα πολύ μικρό μερίδιο της ε, βοήθειας που διανέμεται προς εκείνη την κατεύθυνση. Όπως ξέρετε, η αρρωγή δεν σημαίνει φιλανθρωπία, σημαίνει μόχλευση. Σημαίνει δηλαδή ότι μπορούμε να επηρεάζουμε τους εταίρους μας. Άρα το θέμα είναι καθαρά πολιτικό, δεν είναι χορηγούμε, δεν χορηγούμε βοήθεια. Δεύτερον, ε, ποιο θα, ποια θα είναι η έκβαση, ποια είναι η έκβαση της Ευρώπης, η Ευρώπη θα τα καταφέρει ή θα διαλυθεί. Ε, νομίζω ότι Ίσως η Κίνα σε αυτό ευελπιστεί, αλλά για τη Βραζιλία η Ευρώπη θα βρίσκεται εδώ για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι μια μεγάλη δύναμη. Η Βραζιλία έχει διμερείς ε, σχέσεις με πολλές χώρες μεμονωμένα της Ευρώπης για θέματα τεχνολογίας, εκπαίδευσης, εμπορικών σχέσεων και ούτω καθεξής. Ως προς την εμπορική πολιτική λέγαμε ότι η διαφορά μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήπα στην εμπορική πολιτική είναι ότι η ήπα είναι ένας τίγρης, περικυκλώνει το θύμα ε, και στη συνέχεια αναπηδά και του κόβει ένα κομμάτι. Η Ευρώπη είναι ένας μεγάλος υποπόταμος με ένα μεγάλο μηδίαμα, μικρά ματάκια και μυρικάζει, μυρικάζει, μυρικάζει το όλο ζήτημα και όταν το θύμα δεν κοιτά, τότε κάθεται, επικάθεται στο θύμα της. Έτσι βλέπουμε την Ευρώπη. Ε, και έτσι είδε και η Βραζιλία τον κανονισμό Δηλαδή, οι κανονισμοί σας μπορεί να έχουν καθολική εμβέλεια. Αυτό μπορούσατε να το κάνετε πολύ εύκολα, αλλά τώρα αντιδρούν. Γι' αυτό μίλησα για no regulation without representation. Γι' αυτό νομίζω ότι βρισκόμαστε μαζί στο ίδιο ε, καράβι, αν θέλετε, σε αυτή τη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση. Εάν βουλιάξετε εσείς, θα βουλιάξουμε και εμείς. Και αν οι χώρες BRICS βουλιάξουν, το ίδιο θα κάνει και η Ευρώπη. Τον 20ο αιώνα είχαμε έναν τρόπο αντιμετώπισης του συστημικού αυτού προβλήματος με τον πόλεμο. Δηλαδή σκοτώνουμε πολλούς, καταστρέφουμε το κεφάλαιο και μετά να συντάσσουμε την οικονομία. Σήμερα τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα και ελπίζω να μην ακολουθήσουμε αυτή την οδό. Άρα το μόνο που υπολείπεται είναι η συνεργασία. Και ξέρουμε στην Ευρώπη πώς έχουν τα πράγματα και ως προς τον Πολωνό συνάδελφο ποιος θα έχει ηγετικό ρόλο, κανείς. Κανείς και αυτό είναι το πρόβλημα οι μόνοι ηγέτες θα είναι αυτοί που θα εγγυηθούν τα βασικά δημόσια αγαθά. Και οι μόνοι που το κάνουν μέχρι τώρα είναι είπα, είτε μας αρέσει είτε όχι. Δηλαδή ε, μπορούν να εγγυηθούν αυτά τα ε, κοινά δημόσια αγαθά. Η Ευρώπη δεν το κάνει, η Κίνα, η Βραζιλία και η Ινδία δεν θέλουν να το κάνουν και βρισκόμαστε σε αυτόν τον κύκλο. Ως προς το ερώτημα του κυρίου Βανόρτεν, εμπορική πολιτική και εξωτερική πολιτική. Η εξωτερική πολιτική αφορά το εθνικό συμφέρον, το ευρωπαϊκό συμφέρον. Εάν όμως θέλετε να καταρτήσετε την εξωτερική σας πολιτική με βάση το, το εμπόριο, θα πρέπει να ξέρετε ποια είναι τα συμφέροντά σας. Και όταν προασπίζετε έναν τομέα, μπορεί αυτό να είναι αρνητικό για έναν άλλον. Άρα η εμπορική πολιτική αποτελεί μία ολισθένουσα πολιτική μεγάλων λόμπι ε, υπέρ, υπέρ του προστατευτισμού των μειονοτήτων προστατευτισμού. Η, πολιτική, η εξωτερική πολιτική δεν αποτελούσε κάτι τέτοιο. Τώρα όμως μετατρέπεται σε κάτι τέτοιο. Αν θέλετε να καταρτήσετε μία ε, πολιτική με όλα τα λόμπι να προστρέχουν και να φωνασκούν. Σε, αυτό τον, ε, σε αυτή την ε, αλληλεξάρτηση των ε, αλληλεξαρτώμενο κόσμο, οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι οι εθνικές κυβερνήσεις μπορούν να επιλύσουν όλα αυτά τα μεγάλα θέματα. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε να ε, επανέλθουμε σε αυτό που είπε ο κύριος Λανσμπέρκης. Υπάρχει ένα, δημοκρα... Υπάρχει ένα δημοκρατικό χάσμα. Και ως προς τον κύριο Κέλαμ για την αύξηση του, ε, του κράτους δικαίου οι Κινέζοι, οι Ινδοί, όχι τόσο οι Βραζιλιάνοι γιατί ήταν μέσα στα πράγματα, οι Κινέζοι και οι Ινδοί ε, θεωρούσαν ότι οι κανόνες έγιναν από τους άλλους. Δηλαδή λένε εσείς καταρτήσατε τους κανόνες, ε, θέλετε όμως εμείς να ακολουθήσουμε αυτούς τους κανόνες που καταρτήσατε εσείς. Άρα θα πρέπει να τους δώσουμε μία φωνή, μία δυνατότητα συμμετοχής για να είναι και υπόλογοι και για να έχουν όλο ένα και μεγαλύτερη ε, φωνή, μεγαλύτερο πολιτικό βάρος. Βρισκόμαστε λοιπόν σε δύσκολους καιρούς. Υπάρχει η δυνατότητα να ε, και ελοχεύει μια πραγματική κρίση και ενδεχόμενα και πόλεμος. Δηλαδή το χάος θα μπορούσε να υπερισχύσει εάν δεν παίξουμε σωστά το παιχνίδι. Κατ' εξαίρεση, ο κύριος Σαλαφράγκα έχει το λόγο. Ξέρουμε, ξέρουμε ότι έχει πολλά να πει. Έχετε το λόγο. Ζητώ συγγνώμη γιατί έφτασα καθυστερημένο στη συζήτηση έφτασα από άλλη συνεδρίαση να συγχαρώ τον κύριο Σαρισβόλσκι που οργάνωσε αυτή την ακρόαση να συγχαρώ και όλους τους ομιλητές δυστυχώς ε, δεν κατάφερα να ακούσω την αρχική παρουσίαση του κύριου Βαλιαντάου Το γνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια. Άκουσα και την απάντησή του στις ερωτήσεις. Φαντάζομαι θα ήταν τόσο λαμπρός όσο πάντα. Ε, θα ήθελα να του θέσω το εξή ερώτημα. Φαντάζομαι πως γνωρίζετε μια ενδιαφέρουσα μελέτη του Ινστιτούτου Ελκάνου για την παγκόσμια επίδραση. Σε 35 χρόνια λέγεται ότι ο οικονομικός άξονας θα μετακινηθεί προς τον Ειρηνικό και τον Ινδικό ωκεανό από, από τον Ατλαντικό. Παρ' όλα αυτά αυτή η μελέτη λέει σαφώς ότι η μόνη υπερδύναμη αυτή τη στιγμή, οι Ε, Πολιτείες, είναι τρει φορέ πιο ισχυρή από, τι τέσσερις, επόμενε οικονομικέ δυνάμει, επόμενες οικονομικές δυνάμεις, ε, μεγαλύτερη από την Ιαπωνία και τη Ρωσία κλπ. Ε, και αναφέρεται σε ορισμένα μικρά κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση Λέει ότι η Αυστρία δέχεται δύο φορέ περισσότερους μετανάστε από τη Βραζιλία, η Δανία ξεπερνάει σε υπηρεσίες στη Ρωσία, η Σλοβενία ε, κερδίζει τρεις φορές περισσότερα μετάλλια από την Ινδία σε αθλητικές οργανώσεις και η Ελλάδα ε, από επιστημονικής πλευράς ε, ε, έχει περισσότερες δημοσιεύσεις από την Νοτιοφρική. Βέβαια όλα αυτά θα πρέπει να τα βάλουμε στο σωστό τους πλαίσιο γιατί το σημαντικό είναι οι τάσεις και όχι τα στιγμιότυπα. Και μιλάμε για μερικά μικρά κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μιλούσαμε για τα μεγαλύτερα, ε, βέβαια αυτά τα στοιχεία θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο γλαφυρά. Συνεπώ, με βάση αυτή την πραγματικότητα και δεδομένου ότι εσεί ξέρετε πολύ καλά την ε, Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Μερκοσούρ, ε, συζητάμε μια αναθεώρηση του προπολογισμού του 2011 που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να περικόψει ε, προ προς το Μεξικό και τη Βραζιλία για παράδειγμα για να τους μεταφέρει στη Βόρεια Αφρική και την Μεσόγειο. Πώς εσείς, μα γνωρίζουμε ότι αυτές οι χώρες ε, BRICS δεν χρειάζονται δάνεια, χρειάζονται ε, ευκαιρίες μέσω των συμφωνιών σύνδεσης. Ε, εν πάση περιπτώσει, εσείς αυτές τις περικοπές ε, Πώς τις ε, ερμηνεύετε. Περικοπές από συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές είναι, ε, αποτελούν ένα πολιτικό μήνυμα σε ό,τι αφορά τη σημασία των χωρών BRICS για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ε, πιστεύετε ότι θα έπρεπε να μην περικοπούν αυτές οι συνεισφορές που έτσι κι αλλιώς είναι συμβολικές προς τις χώρες BRICS. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς. Ε, για να απαντήσει τώρα ο καθηγητής Βαλερά. Η ερώτηση είναι δύσκολη και η απάντηση είναι εξίσου δύσκολη. Γιατί αφενός είναι πολύ θετικό το μήνυμα ότι η Ευρώπη αρχίζει να ενδιαφέρεται για το τι συμβαίνει στη Βόρεια Αφρική. Να δούμε, θα είναι πιο σοβαρή στη σχέση της με τις χώρες ε, ε, με τις αραβικές χώρες και τις χώρες του, της Βόρειας Αφρικής ε, που μετά την ε, Αραβική Άνοιξη έχουν πια την δυνατότητα να εξελιχθούν σε κάτι πολύ καλό. Από συμβολικής πλευράς το να έχει κάποια σημασία ε, το ότι μειώνονται οι ε, επιδοτήσει προ τη Βραζιλία και το Μεξικό. Αλλά έτσι κι αλλιώ δεν, δεν τη χρειάζονται αυτή την επιδότηση αυτέ οι χώρε. Αυτό που χρειάζονται είναι περισσότερε ευκαιρίε, περισσότερο εμπόριο, ε, περισσότερα πράγματα από κοινού, κοινού δράση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα στην Αφρική, τριγωνικέ συνεργασίε κλπ. Χιλιάδε πράγματα που μπορούμε να κάνουμε από κοινού. Το πρόβλημα τη Ευρώπη με την Βραζιλία πιο συγκεκριμένα από τις χώρες του Μαρκοσούρ εξακολουθεί να είναι η διαπραγμάτευση Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ. Βλέπουμε ότι οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή ε, μειώνουν τις επιδοτήσεις στην εθανόλη. Για λόγους άσχετους με την εθανόλη όμως. Οπότε οι Βραζιλιάνοι θα συνεχίσουν να παράγουν εθανόλη για τις ε, ε, ενώ η Ευρώπη δεν τους επιτρέπει. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και αυτά τα μηνύματα είναι τα πιο δύσκολα να ερμηνευτούν γιατί η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι έτοιμη να μπει σε μια βαθιά σχέση με τις χώρες της Αμερικής όπως ιδιαίτερα τη Βραζιλία ή όχι. Σε ποιο βαθμό η Ευρώπη συμφωνεί να συμφιλειωθεί με τα συμφέροντα του τη άλλη πλευρά, χωρί να λέει εμεί έχουμε δίκιο και εσεί άδικο. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από τη μείωση ή όχι κάποιων επιδοτήσεων προς τις ε, χώρες αυτές Μεξικό και Βραζιλία. Δεν ξέρω αν καταλάβατε την απάντησή μου. Είναι λίγο δύσκολη η ερώτηση και είναι δύσκολη και η απάντηση. Bene. Καλώς. Ευχαριστώ τους ε, ομιλητές μας και τους ε, συναδέλφους που συνεισέφεραν στο να γίνει ενδιαφέρουσα εκπρόση αυτή και προχωρούμε στο επόμενο θέμα. Σύσταση προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Μολδαβίας. Σας θυμίζω ότι είναι η δεύτερη εξέταση της σύσταση προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή για τις διαπραγματεύσεις της Συμφωνίας Σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μολδαβίας. Σας ενημερώνω ότι έχουν κατατεθεί 92 τροπολογίες εκ των οποίων 9 συμβαστικές τελικά ε, καταθέτει ο εισηγητής. Η Επιτροπή Ίντα ψήφισε ε, σήμερα ε, το μεσημέρι ε, τη γνωμοδότησή της που θα εξετάσουμε αύριο. Αν είναι έτοιμος ο εισηγητής ο κύριος Γότσον θα του δώσω μέσα το λόγο για να μας παρουσιάσει την κατάσταση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είστε έτοιμος, μάλιστα. Θα ήθελα να αρχίσω με ευχαριστίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συνεισέφεραν στη συζήτηση αυτής της έκθεσης με πάρα πολύ χρήσιμες υποδείξεις και προτάσεις, καθώς επίσης και τους σκιώδεις εισηγητές των άλλων πολιτικών ομάδων, με τους οποίους είχα την περασμένη ομάδα μια άκρος ενδιαφέρουσα συνεδρίαση. Ως αποτέλεσμα, καταλήξαμε σε μια σειρά συμβιβαστικών τροπολογιών. Uh, explain, uh, chairman, uh, Μπορεί... Ε, να έχω εξηγήσει και θα εξηγήσω ε, ξανά ότι ε, βασικό μου μέλημα ήταν να προσπαθήσω να βρω όσο γίνεται μεγαλύτερη συνένεση για αυτή την έκθεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μιλούμε για χώρες ε, στη ανατολική μας γειτονία να έχουμε ε, αποφάσεις που να βασίζονται σε ευρύτατη συνένεση για το τι μέλη και να βεβαιωνόμαστε ότι μιλούμε με μία φωνή όταν πρόκειται για τις χώρες αυτές και για τη στάση μας. Ακριβώς αυτό κρύβεται πίσω λοιπόν από τις συμβαστικές τροπολογίες τις οποίες σήμερα καταθέτουμε. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου που ε, γνωμοδότησε και σήμερα την ψήφισε. Ο κ. Ντέβιτ Μάρτιν είναι ο συντάκτης και πρέπει να σας πω ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα με τη γνωμοδότηση αυτή ως εισηγητής απολύτως και θα παρακαλούσα τους συναδέλφους να ε, ενσωματώσουμε τη γνωμοδότηση αυτή στην έκθεσή μας με τον τρόπο που ψηφίστηκε σήμερα. Ε, και τροπολογίε πρόεδρε καλύπτουν πολλές από τις άλλες τροπολογίε των συναδέλφων. Ελπίζω να τις έχετε όλοι στα χέρια σας, δεν χρειάζεται να τις διαβάσω μία προς μία. Επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή αλλαγή, να προτείνω να αλλάξει μία συμβιβαστική μετά από περιττέρω συζήτηση που είχα με τους σκιώδεις ηγητές. Είναι η συμβαστική τροπολογία που καλύπτει την παράγραφο 1α. Ο νέος συμβιβασμός λοιπόν έχει ως εξής. Και ζητώ συγγνώμη γιατί είναι μεγάλη φράση αυτή στα αγγλικά. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να συνεισφέρω και εγώ στην ταχεία ε, εκφύληση της γλώσσας μου. Θα ε, έβαζα πολλά κόμματα εδώ. Γίνεται λόγος για την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θέλω ε, να βάλουμε και όχι την ε, προοπτική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται και συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και βασίζεται αυτό στην αποδοχή ότι η ε, προοπτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 49 της Συνθήκης της Λισαβόνα, θα πρέπει να συμβαδίζει χέρι-χέρι με ε, τις διαθροτικές αλλαγές. Είναι ε, πολύτιμος μοχλός όσο και καταλήτης ε, για την υποστήριξη της κοινή γνώμης στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Και ελπίζω, Πρόεδρε, με αυτή τη μικρή αναδιατύπωση της προτινόμενης συμβαστικής τροπολογίας να βρει τη ευρεία ε, συνένεση των πολιτικών ομάδων και υποστήριξη. Βεβαίως, Πρόεδρε, ευπρόσδεκτα τα σχόλια ή προτάσεις των συναδέλφων. Yes, thank you. I give the floor to the shadow... Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στους και ηγητές. Ο Γκουράνου πρώτος, Τράιον. Yes. Very, no. oh, right here in front. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή ο οποίος ε, κατέδειξε επικοδομητικό πνεύμα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και κατά τη διάρκεια των ζωηρών συζητήσεων. Χαίρομαι διότι έδειξε μεγάλη ευελιξία, είχε υψηλή κρίση και μπορούμε να δεχτούμε το συμβασμό που μόλις ανακοίνωσε. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή αυτή η διατύπωση δεν υπάρχουν άλλα μείζωνα ζητήματα τα οποία ε, μας απασχολούν ως προς τις ε, τροπολογίες. Νομίζω ότι έχουμε υπερβεί τα μεγαλύτερα εμπόδια και θα ήθελα για άλλη μια φορά να πω ότι συμφωνώ σε σχέση με τη φθήνουσα πορεία που ακολουθεί η αγγλική γλώσσα. Ο Ιωάννα Πάσκου αντιπρόεδρος της ε, Επιτροπής ΑΦΕΤ. Έχετε το λόγο. Και εγώ, κατά παράδοξο τρόπο, δεν έχω τίποτα να αντιτάξω σε αυτά που είπε ο κύριος Σουγκουρεάνου για αυτή την έκθεση. Υποστηρίξαμε την άποψη ότι ότι ο εισηγητής ε, έκανε μια πολύ καλή και επαγγελματική εργασία και προσπάθησε να βρει συμβιβασμούς για ορισμένα βασικά στοιχεία. Υποστηρίζουμε λοιπόν και αυτή την αλλαγή της τελευταίας στιγμής που αναφέρθηκε γιατί θέλουμε να γίνει ένα βήμα προς τα εμπρός ως προς τις βασικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να επιτελεστούν στη Μολδαβία για να προσχωρήσει κάποια στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επενδύσαμε πολλά σε αυτή την έκθεση. Έγινε μία εις εργασία και συμφωνώ με αυτά που προείπε ο κύριος Ουγγουράνο ως προς την προσωπική συμμετοχή του εισηγητή για να ε, βρεθεί μια λύση σε αυτό το σημαντικό θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο και τους συναδέλφους για την ε, εμπεριστατωμένη αυτή εργασία. Βέρνερ Σούλτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σιγητά, Καταλήξαμε σε μεγάλη συμφωνία, την οποία επιτύχαμε πραγματικά. Είναι ε, μια έκθεση πάρα πολύ ισόρροπη, ε, που ενθαρρύνει μια πολύ ελπιδοφόρα χώρα και υποστηρίζει τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, τις τονίζει και τις υπογραμμίζει. Και χαίρομαι που στο ένα επίμαχο θέμα που εκκρεμούσε και μόνο ε, καταλήγουμε ε, με μία ευφυή διατύπωση να δώσουμε ένα προσανατολισμό με το συμβιβασμό στο άρθρο 49 και στην ευρωπαϊκή προοπτική. Είμαι πολύ ικανοποιημένο με την έκθεση. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά ειλικρινά τον εισηγητή για την πολύ καλή συνεργασία που ε, κατάφερε να φτάσει σε μια τόσο μεγάλη συμφωνία. Νομίζω ότι θα προχωρήσει η ε, Μολδαβία χάρη στην έκθεση αυτή και νομίζω θα χαροποιήσει και τους πρωταγωνιστές. Και εμείς uh, α, ως ομάδα συμφωνούμε με τον συνάδελφο τον οποίο έχει τιμήσει η ίδια η Βασίλισσα. Νομίζω ότι θα πρέπει να πω προς τους Ρουμάνους συνδελφούς σε σχέση με το θέμα της Μολδαβίας και επειδή ήμουν μέλος για 8 χρόνια, θεωρώ ότι η διατύπωση που χρησιμοποιήθηκε για τη Μολδαβία και την Ουκρανία, που είναι και μεγαλύτερη χώρα, διαφέρει το ε, θέμα αυτό αφορά τις οικονομικές, ε, τις ευρωπαϊκές προοπτικές της χώρας πέρα από την ε, προσέγγιση σε σχέση με το ΝΑΤΟ. Εν πάση περιπτώσει, εάν γίνει μια συζήτηση για την Ουκρανία θα πρέπει να υποστηρίξετε την προοπτική, την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας και ιδιαίτερα ως προς τις χώρες ε, αυτές τις ανατολικής εταιρικής σχέσεις, δηλαδή την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Λευκορωσία. Δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφορετική διατύπωση, διότι αλλάζει το σημασιολογικό πεδίο και αυτό είναι νομίζω λάθος. Ας έχουμε μία λοιπόν ενιαία διατύπωση για όλες αυτές τις χώρες και να μην γίνονται διαφοροποιήσεις οι οποίες δεν έχουν έμπρακτα καμία διαφορά αλλά νομίζω ότι οι Ουκρανολόγοι και οι Μολδοβολόγοι ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Ο κύριος Πάσκου χωρίς μικρόφωνο. Let me say. Collega Salafranca, prego. Ο κύριος Σαλαφράγκα, παρακαλώ. Παρόλο ότι ο σκιώδη συγητής μα, ο κ. Ογκουρεάνο, ε, ε, ε, παρουσίασε τη θέση μας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βάτσον για τη δεκτικότητά του, την διαλεκτικότητά του. είναι ένα θέμα αρκετά ευαίσθητο καταλαβαίνω πολύ καλά την λογική που μας ζητάει ο κύριος Τάνοκ. Δηλαδή να είμαστε συνεπείς σε ό,τι αφορά το σύνολο των βρίσκονται στην ίδια θέση. Η πρόταση του κύριου Βάτσον είναι αποδεκτή και θα την υποστηρίξουμε. Θα υποστηρίξουμε όλη την έκθεση όπως είπε και ο κύριος Ευχαριστώ. Ε... Η κυρία Μακοβέη. Oh, Ευχαριστώ. Καταλαβαίνω ότι συμφωνήσαμε τις προφορικές τροπολογίες του εισηγητή. Αυτό με χαροποιεί. Να πω και δύο λόγια για την αναφορά στο άρθρο 49 της συνθήκης. Το πιο σημαντικό είναι ότι στην περίπτωση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας ε, εξετάζουμε το κατά πόσον αξίζει, αξίζουν τα επιτεύγματά της. Δηλαδή ποια είναι τα επιτεύγματα της κυβέρνησης και του λαού που καταβάλει σημαντικές προσπάθειες με πολύ θετικά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι η τεχνική αξιολόγηση η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην πολιτική μας απόφαση. Συνεπώς, εξετάζουμε μια ακόμα φορά τι έκανε η χώρα, αξιοκρατικά δηλαδή, και αυτό θα πρέπει να αναγνωριστεί και να ενθαρρυνθούν να συνεχίσουν με τις μεταρρυθμίσεις. Γιατί τελικά αυτός είναι ο στόχος μας, να ενθαρρύνουμε και να υποστηρίξουμε τη χώρα να συνεχίσει με ρυθμίσεις της προς όφελος του λαού. Δεύτερο σχόλιο που έχω να κάνω, στις 15 ε, και 16 Ιουνίου έλαβε χώρα η συνεδρίαση ε, στις Βρυξέλλες με τους συναδέλφους από το Κοινοβούλιο της ε, Μολδαβίας. Ε, εκεί υιοθετήσαμε διάφορα ψηφίσματα σχετικά με την ανάπτυξη της χώρας, σας το λέω ενημερωτικά. Οι συστάσεις στάλησαν έτσι και αλλιώς επισήμως στην Επιτροπή. Αφέτο. Rapporteur for the Thank you, Chair. I consider myself to be extremely fortunate to be the Σουάτσον, ε, χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εισηγητή για τη Μολδαβία και όχι ενό από του μεγάλου γειτονέ τη. Ευχαριστώ πολύ του και οδηγητέ ε, για τα καλά του λόγια και για την υπομονή του. Ευχαριστώ επίσης την κυρία Μακοβέη και την αντιπροσωπεία της Πιστεύω ότι η έκθεση αυτή θα εκπέμψει ένα σαφές μήνυμα προς τη Δημοκρατία της Μολδαβίας ότι η, η πρόοδος της μεταρρυθμίσης ε, που επιτελούνται και η πρόοδος στην κατάσταση της υπερδνηστέριας ε, θα συνοδευτούν από αυξημένη υποστήριξη από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, επί τη βάση της αρχής που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταμοιβή των επιτευγμάτων. Ο κύριος ε, ε, Πάσκου είπε ότι ε, η χώρα αυτή είναι μικρή και όμορφη και αυτό έχει πλέον εκτίματα μερικές φορές. Η κυβέρνηση της μέσα σε ένα δύσκολο πλαίσιο κατάφερε να προχωρήσει τη χώρα. Εγώ θαυμάζω την πρόοδο που έχει επιτύχει η Μολδαβία και ελπίζω ότι αυτό θα μας επιτρέψει να συνάψουμε ακόμα πιο στενές σχέσεις με την χώρα. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να ψηφίσουμε αύριο. Ευχαριστούμε συνάδελφε και διακόπτουμε για 10 λεπτά μέχρι τις 5.30 για να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Beh, questo lo vedranno, eh,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

Υπότιτλοι AUTHORWAVE <clears throat> Αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να τηρήσουμε το ωράριό μας και να υποδεχτούμε τον προσκεκλημένο μας. Αρχίζουμε με πολύ μικρή καθυστέρηση σε σχέση με την ημερήσια διάταξη, αλλά κάτι τέτοιο επιβαλόταν για να τον υποδεχτούμε. Δεν θα πρέπει όμως να καθυστερήσουμε περαιτέρω και θα ήθελα να καλωσορίσω τον εκπρόσωπο τύπου του Συμβουλίου Αντιπροσώπων της Δημοκρατίας του Ιράκ για την διερμηνία έχετε το κανάλι 17 για τη διερμηνία προς τα αραβικά. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα διαπιστώνουμε πόσο έχουν ενισχυθεί οι σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοβουλίων. Η Επιτροπή μας ενδιαφέρεται άμεσα για τις δημοκρατικές εξελίξεις στη χώρα σας και αυτό καταδεικνύεται από πολλά γεγονότα που θα απαριθμίσω αποφασίσαμε να αναθέσουμε στον πλέον ικανό συνάδελφο, τον κύριο Μάουρο, που είναι και επικεφαλής της αντιπροσωπείας του κόμματός μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Του αναθέσαμε λοιπόν μία έκθεση για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιράκ. Απεστάλλει μία αντιπροσωπεία με επικεφαλή στον κύριο Στίβενσον, υπεύθυνο της αντιπροσωπείας ε, για τις σχέσεις με τη χώρα σας που συναντήσατε στη Βαγδάτη τον Απρίλιο και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω γιατί βρίσκεται εδώ στο Προεδρείο. Στη συνέχεια διενεργήθηκε μια δημόσια ακρόαση από την Επιτροπή μας τον Μάιο που ασχολήθηκε με την οικονομική και κοινωνική κατάσταση στη χώρα σας. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης εκείνης ακούσαμε πολλές μαρτυρίες που μας συντάραξαν και διαπιστώσαμε τι συμβαίνει, ποιες είναι οι εξελίξεις Πρόκειται για μια κατάσταση που θα πρέπει να οδηγήσει στην ευημερία του Ιράκ για όλους τους ε, πολίτες ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές τους πεπιθήσεις. Θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και ελευθερίας. Σε αυτές τις, ε, ε, στις αξίες σταθήκαμε και θα ήθελα να τονίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αλληλέγγυο και θα ήθελα να σας βοηθήσει σε αυτή τη δύσκολη πορεία σας. Είχαμε και την Συμφωνία Εταιρικής Οικονομικής Σχέσης μεταξύ Ιράκ και Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα εξετάσουμε τους επόμενους μήνες και που θα εγκρίνουμε και πιστεύουμε ότι θα προωθήσει τις διμερείς μας σχέσεις. Το Ιράκ είναι μια πλούσια χώρα, όχι μόνο εξαιτίας των φυσικών της πόρων, αλλά και επειδή έχει μια μεγάλη και μακραίωνη ιστορία και πολιτισμό. Επίσης, ο λαός της χώρας σας έχει ταχθεί υπέρ των ανθρωπίνων ε, αξιών, ήταν ένας λαός αδάμαστος και έχει την ταυτότητά του, την ίδια ταυτότητα την οποία σεβόμαστε. Οι προκλήσεις είναι πολυάριθμες που πρέπει να αντιμετωπιστούν. θα τις συζητήσουμε. Θα ήθελα να καλωσορίσω λοιπόν την αντιπροσωπεία του Ιράκ. Σας δίνω άμεσα το λόγο και θα ήθελα να περιοριστείτε σε 15 λεπτά έτσι ώστε να προωθήσουμε και έναν διάλογο έτσι ώστε να προωθήσουμε αυτή την συνεργασία, την συνεργατική στάση. Σας ευχαριστώ πολύ και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Αλμπερτίνη, Πρόεδρε της Επιτροπής Εξωτερικών. Είναι πολύ καλή ευκαιρία που έχουμε. Θα ήθελα να σας ε, χαιρετήσω εξ ονόματος του ε, Ιρακινού λαού και τους λαούς της Ευρώπης. Σαλάμ, ειρήνη προς όλους και ελπίζω στο μέλλον να έχουμε καλές σχέσεις όλοι οι λαοί ε, με βάση τη ε, συμπάθεια, τη φιλία, την ε, αλληλεγγύη και την υποστήριξη. Να καταλήξουμε σε ένα κόσμο ειρήνης χωρίς πολέμους, χωρίς κρίσεις, σε ένα κόσμο ισότητας και δικαιοσύνης μεταξύ όλων των λαών της γης. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ένα από τα χαρακτηριστικά με τα οποία πρίκυψε ο Θεός, ο το λαό μας είναι ότι ο λαός μας είναι πάρα πολύ ε, ζωντανός και ανθεκτικός. Κάθε φορά που το σαρώνουν καταιγίδε επανέρχεται. Κάθε φορά που καταστρέφεται τη χώρα και η οικονομία ε, σηκώνεται όρθιος ο λαός μας και προσπαθεί να επανέλθει. Όπως ο Φίνικας που ε, φυτρώνει από τις τάχτες του και επανέρχεται δρυμύτερος και από την αρχή η χώρα μας και ο λαός μας πρέπει να πούμε ότι ανήκει στις ε, πρώτους πολιτισμούς της γης, έδωσε τους πρώτους κώδικες και την πρώτη τέχνη, τις πρώτες τέχνες, την πρώτη δημιουργικότητα. Και αυτό που σήμερα είναι κατάρα για το Ιράκ μπορεί στη συνέχεια να γίνει ευλογία. Και ελπίζουμε οι λαοί μας και ο λαός μας να μείνει στο μέλλον ε, πάντα όρθιο. Βεβαίω γνωρίσαμε πάρα πολύ δύσκολου καιρούς και η χώρα και ο λαό. Η χώρα καταστράφηκε, ε, η υποδομή μας επίσης ε, αποκλειστικά. Η κατάσταση είναι ικτρή και ήμασταν πεδίο μαχών και μάλιστα κατεξιοδότηση ορισμένων κρατών που ανέθεταν σε άλλους και πλήρωσε μεγάλο τίμημα ο λαός και οι αθώοι Ιρακινοί. Σήμερα ο λαός του Ιράκ δεν καταλαβαίνει από πού πήγαζαν όλα αυτά τα δεινά του. Έχουμε πολλούς ε, εκτοπισμένους, πολλούς ανθρώπους που έχουν χάσει τις αιστείες τους, ε, πολλές ε, δυνάμεις που συγκρούονται στο εσωτερικό της χώρας, πολλές δυνάμεις που θέλουν να επιδράσουν από το εξωτερικό. Ακούμε διάφορες εκδοχές, ψεύδι πολλά για το τι συμβαίνει στη χώρα κατά κάποιο τρόπο υπάρχει μια φωνή από το εσωτερικό της χώρας που θέλει να την καταστρέψει, να την κατακαιρματίσει, να την χωρίσει και να ε, την κάνει ένα σωρό συντρίμια με πολέμους πραγματικά για όνομα άλλων. Ορισμένοι ε, αξιοποιούν αυτό το, το κενό, συγγνώμη, το εκμεταλλεύονται ε, για να κάνουν ληστείες, ε, λαιλασίες. Η χώρα μας θέλει να ανακτήσει την κυριαρχία της παντού σε όλη την επικράτειά της και να έχει τον έλεγχο και του πλούτου και του μέλλοντός της. Με τη νέα δημοκρατική διαδικασία έχουμε τώρα ένα κοινοβούλιο το οποίο προσπαθεί να είναι η φωνή του λαού για να έχουμε ένα ενωμένο δημοκρατικό Ιράκ που να εγγυάται την ειρήνη και τη σταθερότητα για τους κατοίκους, τους πολίτες. Δυστυχώς όμως όλα αυτά που ελπίζουμε και όλα αυτά που θέλουμε καταραίουν, καταστρέφονται και δεν μεταφράζονται στην πράξη. Η, νεαρή δημοκρατία μας ε, δοκιμάζεται από θρησκευτικές διαμάχες και εμείς ε, ως μέλη του Ιρακινού Κοινοβουλίου προσπαθούμε ε, να είμαστε χρήσιμοι και στο μέλλον θέλουμε να είμαστε ε, πιο ε, χρήσιμοι για το λαό μας και να είμαστε η φωνή του λαού, όχι η φωνή της κυβέρνησης στο Κοινοβούλιο. Ε, ο λαός να καταλάβει ότι έχει ισχύ, να είναι δημιουργικός, να είναι εφευρετικός και αυτά που λέμε για τη δημοκρατία δεν είναι κάτι ξένο για το δικό μας πολιτισμό. Η ιστορία μας η ίδια αποδεικνύει ότι η χώρα μας και ο λαός μας ήταν από τους δημιουργούς της δημοκρατίας ε, στην αρχαιότητα. Και αυτό μας το αφαίρεσαν ε, για τόσο πολύ καιρό που ξεχάσαμε πώς λειτουργεί η δημοκρατία. Και μόνο τους τελευταίους μήνες το Ιράκ έζησε μια νέα κατάσταση. Αποδεικνύει ότι ο λαός είναι φιλιρινικός, θέλει να καταπολεμήσει τον εποτισμό, τη διαφθορά ε, και ε, τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος, τις υπεξαιρέσεις, όλα αυτά τα ε, δεινά που μαστίζουν τη χώρα. Σήμερα πραγματικά διακαώς επιθυμούμε να βγούμε από την πολιτική και οικονομική κρίση που διανύουμε και θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να μας βοηθήσετε για να ξεπεράσουμε την κρίση αυτή και να βρούμε λύσεις στα προβλήματά μας για να επανέλθει η χώρα το ρόλο που διαδραμάτιζε στο παρελθόν για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα υπέρ της ειρήνης, της σταθερότητας στην περιοχή και της ευημερίας. Απευθυνόμαστε λοιπόν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα θεσμικά όργανα και στους λαούς της για να επενδύσουν στην οικονομία μας, στη βιομηχανία μας, στην τεχνολογία, στη χώρα μας, διότι είναι και μια αγορά που ανοίγεται σήμερα με μεγάλες προοπτικές. Και όπως γνωρίζετε όλοι, δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι ε, το Ιράκ κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά του προβλήματα, να επανέλθει στην ειρήνη και ε, στην ευημερία και στη σταθερότητα στην περιοχή. Αν συνεχιστεί η κρίση αυτή θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα είναι πολύ ε, καυτή η περιοχή και μάλιστα ένα ηφαίστειο ενεργεία. Χρειάζεται βοήθεια ο του Ιράκ και υποστήριξη στη δέσμευση και στην προσήλωσή του αυτή. Είναι δίκοπο μαχαίρι η κατάσταση στην περιοχή μας και ε, Ε, μάλλον ε, μπορεί να, να γύρει πλάστικα και προς τις δύο πλευρές. Είτε θα είναι ευλογία για την περιοχή, είτε θα είναι κόλαση. Εμείς, ε, επαναλαμβάνω, υποστηρίζουμε και εκφράζουμε το λαό του Ιράκ και όχι την κυβέρνησή του. θέλουμε να είμαστε συμμέτοχοι στον εκδημοκρατισμό, το συνεχιζόμενο στη χώρα. Είμαστε κατά της συνεχιζόμενης καταστολής θέλουμε και καταπολεμούμε στη χώρα μας και τη διαφθορά και γύρω από αυτή. Αλλά όπως γνωρίζετε αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε κατά της πολιτικής δύο μέτρων και δύο σταθμών που καμιά φορά διαπιστώνουμε στην περιοχή μας να ασκείται. Ο νεποτισμός, ο δεσποτισμός, η καταστολή είναι ενιαία φαινόμενα παντού και ε, όπου και να ισχύουν σε οποιοδήποτε σημείο της γης. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να ε, ζητούμε αλλαγές σε μια χώρα, σε μια περιφέρεια και να τις αρνούμαστε ή να τις αγνοούμε κάπου αλλού ή να επισκιάζονται από άλλα γεγονότα και καταστάσεις. Και δεν θα πρέπει να στρεφόμαστε κατά του λαού ε, μιας χώρας, αλλά μέσω της εμπειρίας του Ιράκ μάθαμε τα ε, πρώτα μας διδάγματα. Ότι οποιαδήποτε μικρή ομάδα ε, που ξεκίνησε ε, το θρησκευτικό πόλεμο στο Ιράκ και τώρα έχει κάνει ζώνη θρησκευτικών αντιπαραθέσεων ε, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει να τα γνωρίζουν όλα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. αν παραγνωρίζουμε τα προβλήματά μας δεν θα λυθούν από μόνα τους ε, και κατευθυνόμαστε ευθεία σε ένα τείχο. Ξέρετε ότι για την επίλυση των προβλημάτων μας τα μόνα μέσα δεν είναι τα όπλα. Πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους ειρηνικούς επίλυσης των προβλημάτων. Πρέπει να επαναλάβω ότι θέλω να σας ευχαριστήσω όλους σας για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δώσετε να σας ενημερώσω για την κατάσταση στο Ιράκ. Ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αρχίζει η συζήτηση. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο ε, Στίβενσον, στον συμπρόεδρο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω για την συνεχή σας ε, φιλοξενία και τις προσκλήσεις της αντιπροσωπείας μας για να μεταβούμε, μάλλον να έρθουμε εδώ, να συμμετάσχουμε στη συνεδρίαση της ε, ΑΦΕΤ. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τον κύριο Νατζέφη, τον ε, πρόεδρο του Συμβουλίου Αντιπροσώπων και τη μεγάλη αντιπροσωπεία, τους δέκα δηλαδή βουλευτές, καθώς και τους συμβούλους. Και θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι ήμουν επικεφαλής μιας μικρής αντιπροσωπείας στη Βαγδάτη τον Απρίλιο φέτος και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη μεγάλη σας, την υψηλή σας φιλοξενία και γιατί μας δώσατε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με τον πρόεδρο Ταλαμπάνη, τον ε, πρωθυπουργό Μπαρζάνη. Συναντήσαμε και εσάς, βεβαίως, κύριε Νατζάφη, καθώς ε, και συναντήκαμε με τον Υπουργό Εξωτερικών τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, πολλούς εκπροσώπους του Συμβουλίου. Γι' αυτό ήταν άκρος ενδιαφέρουσα η συνάντηση. Ορισμένα από τα βασικά σημεία που συζητήσαμε κατά την επίσκεψή μας ήταν η κυβέρνηση Εθνικής Ένωσης. Δηλαδή, δεν είδαμε να έχει διοριστεί η Υπουργός Δικαιοσύνης, Ασφάλειας και Άμυνας επίσης. Δεν έχει διοριστεί κανείς υπεύθυνο για ε, θέματα στρατηγικής πολιτικής επίσης. Οι 19 ε, ρήτρες που έχουν οριστεί δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή και αυτό αποτελεί μεγάλη απογοήτευση για εμάς οι 19 ρήτρε της Συμφωνίας του Ερμπίλ και ελπίζουμε να επιτελεστεί πρόοδος. Ήρθα σε επαφή με εσάς και με μέλη της αντιπροσωπείας σας και πιστεύω ότι έχει επιτελεστεί τουλάχιστον μερική πρόοδος για να ε, φτάσετε σε αυτούς τους διορισμούς που είναι κρίσιμη για να φτάσετε στη σύσταση κυβέρνηση, κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να υπάρχει συγκεντρωτισμός εξουσιών στο πρόσωπο του ε, Πρωθυπουργού, όσο ικανό πρόσωπο και να είναι αυτός. Επίσης, στις Απριλίου έγινε μια μεγάλη σφαγή στον καταβλισμό του Άσραπ και θεωρούμε ότι πρέπει να φτάσουμε σε μια επίλυση και του ζητήματος της ανθρωπιστικής κρίσης, να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε οι 3.400 πρόσφυγες από τον καταβλισμό του ΑΣΡΑΠ να μπορέσουν να μεταβούν στη Νορβηγία, ε, Ελβετία, συγγνώμη, Καναδά και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να βοηθήσουμε και για την εγκατάστασή τους ε, στον Καναδά. Η κυρία Ναβεπίλε από, από την ύπατη ε, αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών έχει αναλάβει να διενεργήσει μία ανεξάρτητη έρευνα την οποία υποστήριξε και η Βαρόνη Άστον, η ύπατη εκπρόσωπος εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διερευνηθεί δηλαδή αυτή η μεγάλη σφαγή και να αποδοθούν ευθύνες. Κατά τη διάρκεια του γεύματος σας μίλησα για μια κοινή επιτροπή ε, μεταξύ της δικής σας, του δικού σας Συμβουλίου ε, Αντιπροσώπων στις 5 και 6 ε, Σεπτεμβρίου για να μιλήσουμε για φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ανανεώσιμες, θέματα γεωργίας, βιομηχανίες, και εκπροσώπους βιομηχανιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κατανοήσουν ότι πρόκειται για μια χώρα με μεγάλες δυνατότητες επενδύσεων. Και ελπίζω η διάσκεψη αυτή, στη διάσκεψη αυτή να συμμετάσχουν και οι πρόεδροι Ταλαμπάνη, ε, Μπαρόζο και Μπούζεκ. καθώς και ο Πρωθυπουργός Ντόναλτ Τάσκ από την ε, Πολωνία. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός να μπορέσει να συμμετάσχει στη διάσκεψη. Έχει μεγάλη σημασία αυτή η εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύω ότι μελλοντικά η οικονομία σας θα μπορέσει να ευημερήσει. Το εύχομαι τουλάχιστον ολόψυχα και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο Στίβενσον, το λόγο έχει ο Μάριο Μάουρο που είναι εισηγητής για θέματα του Ιράκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρισκόμαστε εδώ με εσά και την αντιπροσωπεία σας μετά τη συνάντηση της Βαγδάτης. Εμένα με σημάδεψε η συνάντηση της Βαγδάτης. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ο λαός του Ιράκ το πόσο αγαπά τη ζωή που δυστυχώς ε, τίθεται σε κίνδυνο σε καθημερινή βάση. Αυτό με εξέπληξε. Οι άνθρωποι πεθαίνουν διότι κάθε μέρα μεταβαίνουν στην εργασία τους θέλουν να μεταβούν στη διοίκηση, στα κτίρια της διοίκησης, του κρατικού μηχανισμού, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια. Δηλαδή θέλουν να διατηρήσουν ζωντανό τον κοινωνικό ιστό της χώρας και ζουν σε μια κατάσταση τρόμου. Το γνωρίζουν δε πολύ καλά αυτό και ξέρουν τι κινδύνους διατρέχουν. Έχει μεγάλη λοιπόν σημασία η ισορροπία εκτελεστικού και νομοθετικού σκέλους και θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσο πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε διενέργεια νέων εκλογών από την παρούσα κυβέρνηση. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να κινηθεί καλύτερα μέσω μιας κατανομής εξουσίας και αρμοδιοτήτων που είναι και πιο δίκαιοι και πιο αποκεντρωμένοι. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει μια νέα σταθερότητα της κυβέρνησης και μέσα, μέσω των νέων συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Σαλαφράνκα έχει το λόγο συντονιστής του ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω και εγώ τον πρόεδρο της, ε, του Ιρακινού Κοινοβουλίου. Ε, θέλω να του εκφράσω την αλληλεγγύη μας ε, στον αγώνα του Ιρακινού λαού για ειρήνη, δημοκρατία και εμπέδωση των δημοκρατικών θεσμών τάση είναι τάση ομαλοποίηση ό,τι αφορά την παραγωγή πετρελαίου. Αυτό είναι καλό. Επίση είναι καλό το γεγονό ότι έχει μειωθεί σημαντικά η βία, παρόλο που εξακολουθεί να είναι υπερβολικά ψηλό ε, ο αριθμός των θυμάτων 195 ε, έως 200 θύματα το χρόνο παρόλο, παρόλα αυτά βέβαια παλιότερα είχαμε 4.000 θύματα νεκρούς το μήνα το μήνα εννοώ ε, ε, συμφωνώ με, τα όσα, με ορισμένα από είπε και ο Στίβενσον και να πω τι εννοώ. Ε, υπάρχει ε, ένα θέμα με τους υπουργού Αμήνης και Εσωτερικών και με τις αρμοδιότητές τους. Πώς βλέπετε εσείς και οι συνοδοί σας, τους οποίους επίσης καλωσορίζω, το θέμα αυτό. Δεύτερον, θα ήθελα να εκφράσω την ανησυχία μας για τους, ε, ανθρώπους που ήταν στο, στο Ασράφ. Ε, ήδη εκφράσαμε τις ανησυχίες μας και επισήμως ε, έτσι ώστε να μην ξανασυμβούν τέτοιου δραματικά τραγικά γεγονότα αλλά η συγκεκριμένη ερώτηση που θέλω να σας θέσω είναι η εξής ε, υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και στη χώρα σας για την απόσυρση 46.000 ε, Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην επικράτειά σας μέχρι το τέλος του 2011. Η ερώτηση είναι η εξής. Μπορείτε εσείς να εγγυηθείτε την ασφάλεια του ενέργειου χώρου σας, την ασφάλεια ενεργειακής ε, ε, προμήθειας και διανομής πετρελαίου και πώς θα βλέπατε μια ενδεχόμενη παράταση ε, της διατήρησης στρατευμά, αμερικανικών στρατευμάτων στη χώρα σας. Ε, θα θέλατε να παραταθεί η διαμονή τους μέχρι ότου εξασφαλιστεί πλήρωση ασφάλεια ή θέλετε να αποσυρθούν ε, το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστούμε κύριε Σαλαφράγκα. Η κυρία Μπρέπολς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ να Καλωσορίσω θερμά τον πρόεδρο του Ιρακινού Κοινοβουλίου. Χαίρομαι πάρα πολύ που λέει ξεκάθαρα ότι το Ιράκ είναι προσιλωμένο στην ειρήνη και τη δημοκρατία και κυρίω θέλει να εργαστεί στην κατεύθυνση αυτή. Ο πρόεδρος ήδη αναφέρθηκε σε μια σειρά προβλημάτων ε, που αντιμετωπίζετε με την καταπίεση, την καταστολή και θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις. Ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι γίνεται στο Ιράκ σχετικά. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ελευθεροτυπία και την ελευθερία της έκφρασης. Θα ήθελα να παρακαλώ να μου πει ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου εάν υπάρχουν νομοθετικά μέτρα ή άλλα που να έχουν ληφθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ελευθερία της έκφρασης και ο τύπος να εργάζεται με κάθε ελευθερία. Διότι ακούμε από το Human Rights Watch για παράδειγμα και από άλλους ότι δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά να είναι κανείς δημοσιογράφος στο Ιράκ. Ε, υφίσταται εκφοβισμούς, ένας δημοσιογράφος ε, ε ή απειλές. Επίσης, τι γίνεται με τη θανατική ποινή. Γνωρίζετε ότι ε, είναι από τις χώρες οποίες απαγγέλλεται ε, περισσότερο στον κόσμο, η θενατική χώρα στον κόσμο. Και από τότε που το 2004 εγκαθιδρύθηκε, ε, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία έχουν καταδικαστεί σε θάνατο 300 άνθρωποι. Η Ιρακινή κυβέρνηση πάρα πολύ φιδωλά μας ενημερώνει και ε, καμία χιλιοστή άνθρωποι επίσης Χίλια άνθρωποι περιμένουν να εκτελεστούν στους διαδρόμους του θανάτου. Και αύριο, μάλλον σήμερα το πρωί είχαμε τη συζήτηση στην ε, Υποεπιτροπή Ανθρωπινών Δικαιωμάτων για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εσείς μπορείτε να μας πείτε αν έχει γίνει καμία πρόοδο σε σχέση με την κύρωση ε, του καθεστώτος ε, της Ρώμης σε ό,τι αφορά τελευταίο τη κατάσταση των γυναικών στις ε, χώρα σας. Ε, γνωρίζουμε ότι το θέμα της βίας κατά των γυναικών είναι πολύ ε, σοβαρό και εγκλήματα τιμής και ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών και μέχρι και εμπόριο γίνεται με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση των γυναικών. Μπορείτε να μας πείτε τίποτα για τις δράσεις που ανέλαβε ή αναλαμβάνει το Ιρακινό Κοινοβούλιο από αυτόν. Και ένα τελευταίο. Ε, σε ό,τι αφορά τη Μοσούλη που είναι η τρίτη πόλη σε μέγεθος και κρίσιμη για την επιτυχία ε, και την ασφάλεια της κατάστασης στο Ιράκ. Αν δεν απατώμε, εσείς ο ίδιος κύριε Πρόεδρε, πολύ πρόσφατα προτείνατε να ιδρυθεί μια ημιαυτόνομη σουνητική περιοχή στη Μοσούλη, κάτι ανάλογο με το Ιρακινό Κουρδιστάν. Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγο περισσότερο πώς βλέπετε και την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Μπρέπολς. Ο κύριος Άτκινς έχει το λόγο. Uh- ε, καλώς ήρθατε κύριε Πρόεδρε, σε εσά και στα υπόλοιπα μέλη του Κοινοβουλίου. Εγώ νόμιζα ότι ήταν δύσκολο να είσαι κανεί μέλο του Κοινοβουλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, <laughs> αλλά σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολο από το να είσαι μέλο του Κοινοβουλίου στο Ιράκ. Τα συγχαρητήριά μου λοιπόν. Συμπάσχω μαζί σα και κατανοώ πολύ τη γενναιότητά σα. Ε, δύο-τρία σχόλια έχω να κάνω. Πρώτον, δεν φαίνεται να είστε και πολύ θετικό. Διότι ο αριθμός των κομμάτων που βρίσκονται στο Κοινοβούλιο και οι διαφορές τους δεν επιτρέπουν την εύκολη εξασφάλιση ενότητας. Η αντιπολίτευση είναι πάντοτε σημαντική σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, αλλά ταυτόχρονα αν όλοι ε, τα βάζουν με όλους υπόλοιπους δεν είναι εύκολο να προχωρήσει η χώρα. Οπότε Ε, τι ποσοστό των μελών του Κοινοβουλίου υποστηρίζει αυτή τη πράξη κυβέρνηση ε, και πώς είναι αυτοί που αντιδρούν. Δεύτερον, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς εδώ, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να σας βοηθήσουμε. Μπορούμε να ενθαρρύνουμε, μπορούμε να λέμε τα σωστά πράγματα, αλλά υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο που μπορούμε να κάνουμε για να σας βοηθήσουμε. Τέλος, έχω επισκεφθεί την Μέση Ανατολή πολλές φορές τα τελευταία χρόνια και ε, ο πολιτισμός σας έχει επηρεαστεί πολύ από τον, ε, τους πολέμους στη Μέση, Ανατολή ε, και τα αρχαία έχουν πληγεί, έχουν υποστεί πολλές βλάβες επανειλημμένως. Τι έχετε κάνει για ε, να ε, τα επιδιορθώσετε ή να τα ανακτήσετε. Ευχαριστούμε τον κύριο Άτκινς. Ο κύριος Κέλαμ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, εκτιμούμε την παρουσία σας εδώ, τη δική σας και της αντιπροσωπείας σας. Πολλοί συνάδελφοι μας είπαν ότι υπό τις παρούσες συνθήκες το Ιρακινό Κοινοβούλιο αποτελεί μια ζωηρή πηγή ε, δημοκρατίας, ελπίδας και ζωηρής δραστηριότητας. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες για πολιτικο-οικονομικές σχέσεις και όπως ακούσατε ενδιαφερόμαστε άμεσα να αναπτύξουμε αυτές τις σχέσεις. Θεωρείτε ότι η αντιπροσωπεία μας είναι επαρκής. Αναμένετε πρωτοβουλίες ή δραστηριότητες από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο εγγύς μέλλον. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Στίβενσον και με άλλους που ανέφεραν ότι είναι πολύ σημαντικό να συγκροτηθεί η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας στο Ιράκ. Γιατί χρειαζόμαστε έναν αξιόπιστο και αποτελεσματικό εταίρο. Επίσης, στον καταβλισμό Ασράφ, η κατάσταση ήταν άκρος ανησυχητική με τα όσα συνέβησαν θα ήθελα να ρωτήσω πώς ε, αντιμετωπίστηκε η κατάσταση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε πολλά ψηφίσματα για την ασφάλεια αυτών των ανθρώπων στον καταβλισμό. Δηλαδή πρόκειται για μια μεγάλη δοκιμή για την επικράτηση του δικαίου στο Ιρακινό κράτος και επίσης θα πρέπει να χορηγηθεί και ιατρική βοήθεια προς τους τραυματίες και όλους όσους έχουν πληγεί. Ευχαριστούμε κύριε Κέλλαμ. Μπέλτερ. Εκπρόσωπος με τη σχέση στο Ισραήλ και επίσης συζητητής σε μία έκθεση για το Ιράν. Πρόεδρος Εντοπροσωπείας για το Ισραήλ. Ε, ευχαριστώ. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Κύριε Πρόεδρε του Ιρακινού Κοινοβουλίου, καλώς ορίσατε θερμά στο Κοινοβούλιο. Συναντηθήκαμε και κατά τη διάρκεια του γεύματος. Θα μπορούσατε να μας ενημερώσατε ε, για το βαθμό τον οποίο καταλαμβάνει η επιρροή του Ιράν στη χώρα σας. Ανησυχούμε πάρα πολύ για την επιρροή του Ιράν στο Ιράκ. Τι γίνεται με την εθνική κυριαρχία. Eh, και κατάλαβα ότι υπάρχει και ένα θέμα πολιτικού διχασμού. Ποια είναι λοιπόν η επιρροή του Ιράν και μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι ε, υπάρχει και μια οικονομική διαπάλη ε, με την Τουρκία αντίπαλο. Δηλαδή είστε σε μια μέγενη. Από τη μια το Ιράν, από την άλλη η Τουρκία. Πώς έχει η κατάσταση εκεί και η σημαντικότερη ερώτησή μου στη χώρα μου αλλά και εδώ στο Κοινοβούλιο ανησυχούμε πολύ για την ε, πολύ άσχημη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι χριστιανοί του Ιράκ και άλλες ε, θρησκευτικές μειονότητες ε, που υποφέρουν πολύ. Τι κάνει λοιπόν το Κοινοβούλιο από τη δική σας ηγεσία για να προστατεύει τις μειονότητες και να τις κρατάει και στο Ιρακινή επικράτεια. Γιατί το περασμένο μήνα ε, υπήρχε ένας προβληματισμός ε, εμπειρογνωμών και ειδικών που ρωτούσαν υπάρχει μέλλον για τους χριστιανούς στη Μεσοποταμία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπέλντερ. Ε, έχει λήξει η συζήτηση και σας δίνω το λόγο κύριε Πρόεδρε για να απαντήσετε. Shukran jazilan. كثير من الأسئلة متشابهة وأنا سأجيب Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις που έγιναν. Σημείωσα τις ερωτήσεις αυτές. Ο κύριος Στίβενσον ουσιαστικά ε, μιλεί για την εθνική ενότητα και ρωτά τι γίνεται με την εθνική ενότητα και με τους διορισμούς βασικών υπουργών Εθνικής Ασφάλειας, Δικαιοσύνης, Εθνικής Αμήνης και τον καταμερισμό των εξουσιών. Η κυβέρνηση βασίζεται ε, στην πολιτική ε, συνένεση και είναι συνασπισμό όλων των κομμάτων που κέρδισαν τις εκλογές και η συμφωνία αυτή ονομάστηκε Συμφωνία του Ερμπίλ και έχει ρήτρε που μιλούν για μεταρρύθμιση στην εκτελεστική, στην νομοθετική και στη δικαστική εξουσία. Έχουμε διάκριση των εξουσιών στη χώρα. Και επίσης ορίζεται ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία βάσει του εκλογικού αποτελέσματος. Βεβαίως, ε, εφαρμόζεται αυτή η συμφωνία, όχι πλήρως βεβαίως, ε, έχετε δίκιο. Υπάρχουν διάφορες απόψεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η συμφωνία του Ερμπίλ. Βεβαίως υπάρχει καθυστέρηση και πολύ σημαντική στην κάλυψη των Υπουργείων που συνδέονται με την ασφάλεια είναι πολύ δύσκολη η καιρή και όλοι είμαστε απογοητευμένοι. Αλλά μόλις χτες, πριν από τρεις μέρες, ε, έγινε μια συνεδρίαση στο Ιράκ με συμφωνία ε, για εφαρμογή ακριβώς τη συμφωνία του Ερμπίλ εντός ε, δύο εβδομάδων. Και η Επιτροπή Ad hoc δημιουργήθηκε για να συζητηθούν και άλλες ρήτρε και να κάνει συστάσεις για να βγούμε από την κρίση αυτή. Ελπίζω το επόμενο διάστημα, τις επόμενες 15 μέρες, να οριστούν αυτοί οι υπουργοί και να εφαρμοστεί και ε, ο κορμός της συμφωνίας του Ερμπίλ και να υπάρξει και ένας οδικός χάρτης. Αυτό πιστεύω να εφαρμοστεί και άλλωστε εκεί θα δοκιμαστεί και η Ιρακινή Δημοκρατία ε, και το Κοινοβούλιο της χώρας κατά πόσο έχει τη γνήσια βούληση να πετύχουμε και ελπίζω να πετύχουμε. Προβλήματα υπάρχουν όπως και διαφορές άλλωστε, αλλά πιστεύουμε ότι ε, υπάρχει κάποιο ίχνος ελπίδας για να λυθούν. Έρχομαι τώρα στον καταβλισμό του Ασράφ και τα όσα πρόσφατα συνέβησαν. Ε, σαφώς ο καταβλισμός αυτός είναι παλιός καταβλισμός στο Ιράκ και υπήρξαν προβλήματα μεταξύ των όσων διαμένουν εκεί και της Ιρακινής κυβέρνησης και το Κοινοβούλιο δεν δέχτηκε να χρησιμοποιηθεί κανένα είδου βία κατά των προσφύγων εντό της Ιρακινή επικράτεια. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να τιμήσουμε και να αποτίσουμε σεβασμό, μάλλον να σεβόμαστε τους νόμους της χώρας. Ξέρω ότι ε, θανατώθηκαν κάποιοι άνθρωποι νεκρούς ε, στο καταβλισμό του Άσραφ. Ε, χρειάζεται ερευνητική εξεταστική επιτροπή για να δούμε πραγματικά τι έγινε. Ε, το Κοινοβούλιο του Ιράκ θέλει να βρεθεί μια τρίτη χώρα για να υποδεχθεί και να επανεγκαταστήσει τους πρόσφυγες ε, του Ασράφ και ελπίζω πολύ σύντομα να επιλεγεί αυτή η χώρα χωρίς περαιτέρω ε, καθυστερήσεις γιατί είναι ένα θέμα ανθρωπιστικό και διαφέρει όλα τα μέρη. Το σύντομότερο θα πρέπει να επαναγκατασταθούν αλλού εκτός του Ιράκ. Αν είναι πρόθυμη η Ευρώπη να τους δεχθεί στους κόλπους της, αυτή θα ήταν μια λογική λύση σε αυτό το ακαθόδες ε, ζήτημα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ομιλούν ακόμα για επανεγκατάστασή του σε άλλη περιοχή εντός του Ιράκ. Αυτό το απορρίπτουν κατηγορηματικά τα πολιτικά κόμματα. Εμείς λέμε να επαναγκατασταθούν αλλού, σε τρίτη χώρα εκτός του Ιράκ. Έτσι έχει λοιπόν η κατάσταση και προσπαθούμε να ε, την προωθήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Ελπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα να εδρεωθούν αν υπήρξε κάποια κακή συμπεριφορά, ανάρμοστη, λυπούμαστε πολύ. Ε, ε, ε, σε ό,τι αφορά τώρα την εταιρική σχέση με την Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντική και για την Ευρώπη και για μας. Το Ιράκ είναι μια σημαντική χώρα, έχει και πλούτο, έχει και πηγές πλουτοπαραγωγικές και μπορεί να ε, παίξει σπουδαίο ρόλο στη Μέση Ανατολή. Και είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης να συνεργαστεί στενά με το Ιράκ. Τώρα διανύουμε μια μεταβατική περίοδο, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση εντός του Ιράκ και να προωθήσουμε τη δημοκρατία και να εδραιώσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο στη μεταβατική περίοδο από μια ε, αυταρχική κυβέρνηση, από ένα αυταρχικό καθεστώς σε μια δημοκρατική κυβέρνηση. Χρειάζεται να μας δοθεί ευκαιρία να εδραιώσουμε ή να βάλουμε τα θεμέλια ε, και να ε, ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για τις δημοκρατικές αρχές. Ο κόσμος στο Ιράκ είχε συνηθίσει τη βία και την καταστολή. Τώρα θα πρέπει να μάθει πώς λειτουργούν ε, οι νέες ε, καταστάσεις, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στις παλιές αξίες και τις καινούργιες, ότι μπορεί να υπάρξει και κάτι άλλο. Αυτό θα πρέπει να το χωνέψει, να το καταλάβει ο κόσμος και σας χρειαζόμαστε να μας βοηθήσετε ακριβώς με ε, την εταιρική μας σχέση στην αναδιάρθρωση, ανοικοδόμηση της χώρας με επενδύσεις, διότι η ανοικοδόμηση είναι πολύ μεγάλη υπόθεση στο Ιράκ και θα είναι προς αμοιβαίο όφελος όλων των ενεχομένων και των ενδιαφερομένων και εσάς. Απαντώ τώρα στον κύριο Μάουρο, ο οποίος εξέφρασε κάποιους φόβους σχετικά με τις εξελίξεις στο Ιράκ. Εγώ είπα ότι η κατάσταση όντως ε, μας ανησυχεί σοβαρά. Υπάρχουν όμως και μεγάλες προσδοκίες για το τι πρόκειται να ε, ε, έχουμε ως εξελίξεις στο προσεχές μέλλον. Εγώ θέλω να ενεργοποιήσουμε την εταιρική σχέση, να εφαρμοστεί πλήρως η συμφωνία του Ερμπίλ με τους υπουργούς ε, στα χαρτοφυλάκια τους για να καταλάβει ο κόσμος, να έχει μια ωραία εικόνα για το Ιράκ, να δει ότι έχουμε μια κοινή βούληση, να είμαστε πρωταγωνιστές ή, εν πάση περιπτώσει, ενεργοί ε, στα παγκόσμια ε, τεκτενόμενα. Χρειάζονται προσπάθειες και η Βουλή μας είναι πρόθυμη να βάλει τα θεμέλια της δημοκρατίας και να λειτουργεί σωστά. Ο κύριος Τσαλαφράνκα μίλησε επίσης και για την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ε, γνωρίζετε ότι έχουμε 15% της παγκόσμιας παραγωγής ως αποθέματα πετρελαίου. Ελπίζω το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες και έτη, να αυξήσουμε την παραγωγή και να παράγουμε 6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Αυτό είναι στον οδικό μας χάρτη, στα σχέδιά μας και ελπίζω να είμαστε σε θέση να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο την παραγωγή. Χρειαζόμαστε βεβαίως εταίρους για να χρησιμοποιούμε αυτή την ενέργεια του φυσικού αερίου και του πετρελαίου στο Ιράκ. Βεβαίως ε, θέλουμε και είμαστε πρόθυμοι να προμηθεύουμε και την Ευρώπη με ε, φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Υπάρχουν ε, κάποιοι φορείς που σήμερα εκμεταλλεύονται πετρελαιοπηγές ε, στο Ιράκ με μεγάλο δυναμικό και μεγάλες δυνατότητες και ελπίζουμε το Ιράκ να καλύψει το 50% των αναγκών σας τα επόμενα έτη, των ενεργειακών. Κάτι άλλο που είπε επίσης ο κύριος Μάουρο για την κατάσταση που επικρατεί. Ο απότερος στόχος είναι η εταιρική σχέση και θα πρέπει να ενεργοποιηθεί. Είμαστε υποχρεωμένοι να πετύχουμε. Εδώ δεν χωράει καμία αμφιβολία. Ε, πρέπει οπωσδήποτε να πετύχει η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Αν αυτή αποτύχει, τότε προφανώς ανοίγει ο δρόμο για εκλογέ, πάλι θα πρέπει να προσφύγουμε στο λαό ή να ζητήσουμε δημοψήφισμα για να ζητήσουμε τι θέλει ο λαό. Ελπίζω λοιπόν αυτή η εταιρική σχέση να πετύχει, να ορθοποδήσει. Ε, υπάρχουν και άλλα μέσα ε, να συνεργαστούμε και ελπίζω να εφαρμόσουμε, όπως σας είπα και προηγουμένως, τη συμφωνία του Ερμπίλ. Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία ε, για την ασφάλεια με τους Αμερικανούς, όντως λίγοι στα τέλη του έτους. Γινόταν λόγος για 50.000 ε, Αμερικανούς στρατιώτες που θα ανέμεναν στο Ιράκ σε συνεργασία και συντονισμό με τις ε, ε, Ιρακινές αρχές και την κυβέρνηση. Προσπαθούμε να αναθεωρήσουμε τώρα την κατάσταση αυτή της παρουσίας Αμερικανικών στρατευμάτων, αλλά αυτό είναι στα χέρια των ειδικών, των στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων και τον τελευταίο λόγο έχει ο Πρωθυπουργός. Περιμένουμε μια έκθεση που θα κατατεθεί στο Κοινοβούλιο για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα με περισσότερες διευκρινήσεις και ε, σε σχέση με τις ανάγκες, ποιες είναι οι ανάγκες, σε ποιο βαθμό, πώς οι στρατιώτες χρειάζεται να παραμείνουν. Και ε, θα είναι ε, πάντα σε συνάρτηση με τις συνεχιζόμενες απειλές. Η έκθεση αυτή σας είπα θα κατετεθεί στο Κοινοβούλιο, το οποίο θα τη μελετήσει και θα δούμε τι λέει και η κυβέρνηση, γιατί είναι πολιτικό συνασπισμός, ε, απαρτίζεται τα πολιτικά κόμματα. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι η τεχνική αξιολόγηση, εκτίμηση αν χρειάζεται να παραμείνει η στρατιωτική παρουσία των Αμερικανών. θα πρέπει να φροντίσει η κυβέρνηση να μπορούμε να βασιζόμαστε στις ίδιες μας τις δυνάμεις, να είμαστε πιο αυτόνομοι, αλλά να μπορούμε να προσβλέπουμε και στους φίλους μας ε, να ενισχύουμε την κυριαρχία μας. Το επόμενο δίμηνο νομίζω η κατάσταση αυτή θα ξεκαθαριστεί και θα έχουμε και την έκθεση που θα δημοσιεύσει ο, ο Πρωθυπουργό και θα ε, μάθουμε κι εμείς τη φρονεί για αυτά τα θέματα και ειδικά αυτό το τόσο ακαθόδε ζήτημα. Η κυρία Μπρέπουλς για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθεροτυπία και την ελευθερία της έκφρασης γνώμης. Ε, το Σύνταγμα του Ιράκ ορίζει και είναι κατοχυρωμένο στο Σύνταγμα ότι ισχύουν ε, αυτές οι αρχές και τα θεμελιώδη δικαιώματα και η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία της πίστης και ε, βέβαια το θέμα είναι πώς εφαρμόζονται. Η κατάσταση δεν είναι ιδεώδης. Υπάρχουν κάποιες βίες ε, καταστάσεις και υφέρπει η βία πολλές φορές σε μερικά σημεία της χώρας με κακομεταχείριση κρατουμένων που βεβαίως αυτό είναι παραβίαση διεθνών συνθήκων αλλά προσπαθούμε να τηρήσουμε τους νόμους και η κυβέρνηση με την ε, Ιρακινή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρέπει να ορίσουμε τα μέλη της Επιτροπής αυτής που ε, παρακολουθούν και ελέγχουν ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράκ. για να διορθωθούν τα κακό κείμενα και οι κακές συμπεριφορές. Προσεχώς θα οριστούν αυτά τα μέλη και θα εργάζονται όσο γίνεται με πιο ουδέτερο και αντικειμενικό τρόπο και αυτή τη στιγμή συσταθεί λοιπόν η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα μπορέσει να αρχίσει τις εργασίες της. Είναι γεγονός ότι ε, παρατηρούνται κάποιες ε, παραβιάσεις Ο ρεκινός λαός αρνείται αυτά τα φαινόμενα και ε, στρέφεται εναντίον τους και προσβεύει την τήρηση του Ιρακινού συντάγματος. Ελπίζω προσεχώς να αναλάβει τις εργασίες της Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σε ό,τι αφορά την ελευθερία του τύπου είναι σημαντικό. Έχουμε ένα νομοθέτημα για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Είναι νομοσχέδιο αυτό τον καιρό, δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, θα ψηφιστεί στους επόμενους μήνες και θα ε, γίνει νόμος του κράτους για να προστατεύεται η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία ε, λόγου και οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωση θα προστατεύονται και η κυριότητά τους θα γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους και οι ίδιοι θα τυχάνουν σεβασμού και προστασίας. Σε συνεργασία με τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, ε, τως ε, συλλόγους, τι ενώσεις των δημοσιογράφων και άλλους ενδιαφερομένους. Γίνονται πολλές συνεδριάσεις ε, στο Κοινοβούλιο για να είναι σωστός αυτός ο νόμος, διότι ξέρετε ότι ο τύπος είναι η τέταρτη εξουσία. Για τη θανατική ποινή. Είναι ενισχύει ο νόμος αυτός. Έτσι έχει το νομικό πλαίσιο. Προβλέπεται η θανατική ποινή. Αλλά αυτό συμβαίνει μόνο μετά από μία σειρά Ε, διώξεων και ε, αφού, αφού εξαντληθεί ε, κάθε ένδικο μέσο, δικαστήριο, εφετείο, άριος πάγος, ακυρωτικά κτλ. Τελικά εναπόκειται στον πρόεδρο εάν συμφωνεί με τη θανατική ποινή. Όπως γνωρίζετε, η τρομοκρατία προκάλεσε πάρα πολλά θώα θύματα, χιλιάδες στο Ιράκ, με φρικτές ε, δολοφονίες και κάπως θα πρέπει να έχουμε και ένα τρόπο ε, να προστατεύεται η κοινωνία ε, μια αποτροπή απέναντι σε αυτούς τους ανελαίτους τρομοκράτες. Η κυβέρνηση δεν κατέληξε στη θανατική ποινή, ούτε επιβάλλει τη θανατική ποινή ε, κατόπιν ενό απλού αιτήματο. Ε, εξαντλούνται, σα είπα, όλα τα στάδια, όλες οι βαθμίδες της δικαιοσύνης μέχρι να φτάσει στον πρόεδρο. Ο πρόεδρος μου είπε ο ίδιος ότι δεν υπογράφει προεδρικό διάταγμα ε, εκτέλεσης, ναι, αλλά υπάρχουν ε, διαδικασίες και ασφαλιστικές δικλείδες και πάντα κατά περίπτωση. Όταν είναι η δεχθή τα ε, εγκλήματα, οι δολοφονίες, τρομοκρατικές επιθέσεις, η ε, δεχθή, επαναλαμβάνω, λαμβάνουν υπόψη όλα τα στοιχεία για να δούμε αν θα επιβληθεί και αν εφαρμόζεται η θανατική ποινή. Και ελπίζω το μέλλον να είναι πιο λαμπρό στο Ιράκ. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς το Ιρακινό Σύνταγμα προωθεί και προασπίζει και τα δικαιώματα των γυναικών. Προσπαθούμε το 25% των βουλευτών να είναι γυναίκες. Υπάρχει αυτή η ποσόστοση και τώρα την τηρούμε, έτσι ώστε να υπάρχουν ίσοι όροι πρόσβασης στην πολιτική και για τις γυναίκες. Αυτό ισχύει ε, γενικότερα και σε όλα τα συμβούλια, στο Κοινοβούλιο Μιλάμε για ποσόστοση των γυναικών που ανέρχεται στο 25%. Πρόκειται για μία νοοτροπία η οποία ισχύει πλέον στο Ιράκ, δηλαδή προσπαθούμε να προωθήσουμε τα δικαιώματα των γυναικών, να αντιταχθούμε σε μία νοοτροπία σκοταδισμού και αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες έτσι ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν στο κοινωνικό γίγνεσθε. Όλα αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν με ακρίβεια. Όμως διανύουμε μία μεταβατική περίοδο, είναι ε, μεταβατική κυβέρνηση και θα αλλάξουν τα πράγματα πιστεύω στο εγγύς μέλλον. Τώρα, ως προς το ερώτημα... Ως προς το θέμα της Μοσούλης, που θεωρηθεί, θα θεωρηθεί η μη αυτόνομη περιοχή με πλειοψηφία Σουνιτών, προσπαθούμε να προωθήσουμε μία αποκέντρωση, μία διαδικασία αποκέντρωση στο Ιράκ και προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί και έχουν καταβληθεί μεγάλες προσπάθειες. Δυστυχώς όμως ε, έχει αρθεί κάθε δυνατότητα δράσης σε αυτές τις ημιαυτόνομες κυβερνήσεις. Γι' αυτό αυτό που έχει σημασία είναι να προωθήσουμε αυτά τα δικαιώματα των γυναικών και βεβαίως αυτών των ημιαυτόνομων περιοχών. Θα πρέπει να χορηγηθεί αυτονομία σε αυτές τις περιοχές και να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι δεν υπάρχει ούτε μία περιφέρεια η οποία να έχει ένα θρήσκευμα ή μία εθνότητα. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν επαρκώς υπόψη. Δεν θα πρέπει να προβαίνουμε σε σύσταση περιοχών ή αυτόνομων περιοχών με βάση το ε, θρήσκευμα. Μου ελέγχθη επίσης, μου είπε ο κύριος Άτκινς, ότι δεν είμαι αισιόδοξο ως προς την εξέλιξη του πολιτεύματος. Όμως, όπως κάθε φίλη ειρηνιστής, πιστεύω ότι θα επικρατήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα υπάρξει συνένεση, αλλά δυστυχώς κινούμαστε από ένα δεσποτικό καθεστώς, ένα ολοκληρωτικό καθεστώς σε ένα δημοκρατικό. Υπάρχουν πολλά προσκόμματα τα οποία πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να άρουμε. Βεβαίως δεν είμαι ικανοποιημένος, αλλά είμαι αισιόδοξο ως προς το μέλλον της κοινωνίας του Ιράκ. Το κοινοβούλιο μας έχει τρία μεγάλα μπλοκ, τρία μεγάλα κόμματα αλλά και μικρότερα που συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα μεταξύ αυτών των μπλοκ συνεργασίας και γι' αυτό πολλά από τα στοιχεία αυτά δεν έχουν, από τα θετικά στοιχεία που προβάλλουν δεν έχουν πραγματοθεί. Τώρα είμαστε πεπισμένοι ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί η συμφωνία στο σύνολό της. Εμείς ως Ιρακινοί αποζητούμε τη συνεργασία με όλες τις δυνάμεις ειρήνης της Ευρώπης να προωθήσουμε τη συνεργασία, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και θέματα ασφάλειας. Όλοι οι τομείς συνεργασίας παραμένουν ανοιχτοί και εμείς ενδιαφερόμαστε και προσβλέπουμε προς τους Ευρωπαίους φίλους μας. Θα θέλουμε να προωθήσουμε σχέσεις φιλίας και οι Ιρακινοί κάνουν έκκληση προς εσάς για να διαδραματίσετε σημαντικό ρόλο για την ανοικοδόμηση του Ιράκ ως προς ε, θέματα εθνικής κυριαρχίας. Βεβαίως ε, τα έργα τέχνης μας επαπειλούνται. Έχει γίνει κακή χρήση και έχουν καταστραφεί πολλά έργα τέχνης. Πολλά θωρακισμένα βομβάρδισαν συγκεκριμένους αρχαιολογικούς χώρους. Και αυτό δημιούργησε μεγάλες καταστροφές. Ε, μένω ενεός όταν μιλώ για τέτοια ανοσιουργήματα. Επίσης έχουν γίνει πολλές κλοπές. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόγραμμα από το Υπουργείο Τουρισμού να επανέλθουμε επί του θέματος, να αποκαταστήσουμε τα έργα τέχνης και χρειαζόμαστε τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας έτσι ώστε να ασχοληθούμε εκ νέου και με τα έργα τέχνης. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι απάντησα στις ε, περισσότερες ερωτήσεις ως προς την αντιπροσωπεία μας αναφέρθηκε ότι υπάρχει σωστή εκπροσώπηση ότι λειτουργεί πολύ καλά η αντιπροσωπεία σας στο Ιράκ. Θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτούς τους δεσμούς έτσι ώστε να έχουμε μία ενοποιημένη στάση και συνένεση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Θεωρούμε ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Ως προς το χριστιανισμό, οι μειονότητες στο Ιράκ πραγματικά έχουν πληγεί από θέματα θρησκευτικής μυσαλλοδοξίας. Πολλοί Ιρακινοί έχουν πληρώσει αυτή την αδιαλαξία με τη ζωή τους. Πολλές μειονότητες επλήγησαν. Αυτό αφορά μειονότητες αλλά και ολόκληρο τον Ιρακινό πληθυσμό που έχει διωχθεί. Προσπαθούμε να ρίξουμε φως σε θέματα που απασχολούν τις μειονότητες ως προς θέματα κακομεταχείρισης μειονοτήτων και ούτω καθεξής. Θέλουμε οι χριστιανοί να παραμείνουν στο Ιράκ και όχι να απομακρυνθούν. Διότι μιλάμε για μια χώρα που δεν είναι υπέρ της θρησκευτικής αδιαλαξίας. Θα προστατεύσουμε και τις εκκλησίες των χριστιανών. Υπάρχει θέμα διασύνδεσης και με άλλες μειονότητες. γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κατά τη δεκαετία του 20 είχαμε και υπουργού από την μειονότητα των χριστιανών. Γι' αυτό θα πρέπει να τους υποστηρίξουμε ως κυβέρνηση και ως κοινοβούλιο. Και αυτό θα πρέπει να ισχύσει και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πρέπει να δεχτούμε τον εκτοπισμό των χριστιανών. Δεν πρέπει να απομακρυνθούν από τη χώρα προέλευσής τους. Δεν θα πρέπει να δεχτούμε αυτή την τάση. Οι χριστιανοί θα πρέπει να παραμείνουν στο Ιράκ και να διαθέτουν τους ελάχιστους όρους διαβίωσης, εργασίας έτσι ώστε να ενισχυθούν οι θετικοί δεσμοί με, τη... με τα άλλα θρησκεύματα. Αυτό το συζητήσαμε και έγιναν πολλές συστάσεις. Συμφωνήσαμε λοιπόν να συσταθεί μια στρατιωτική δύναμη από τη μειονότητα αυτή των ε, χριστιανών και να υπάρξει και ένα ειδικό ταμείο για να καταβληθούν αποζημιώσεις τους χριστιανούς και να μπορέσουν να οικοδομήσουν τα σπίτια τους και ούτω καθεξής. Έτσι ώστε όσοι επανέλθουν όταν επανέλθουν οι εκτοπισθέντες να μπορέσουν να ζήσουν στα σπίτια τους. Έχει συσταθεί λοιπόν μια επιτροπή ad hoc για να εφαρμόσει τις συστάσεις. Και τώρα διαπραγματευόμαστε αυτό το σχήμα έτσι ώστε να υπάρχει συνεργασία και οι εκτοπισθέντες χριστιανοί να επανέλθουν είναι μεγάλο σφάλμα, είναι εγκληματικό να απομακρύνουμε τους χριστιανούς από την αιστεία τους. Είναι κάτι που δεν είναι αποδεκτό από εμάς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο. Ήταν άκρος ενδιαφέρουσα αυτή η ανταλλαγή απόψεων, αυτή η συνάντηση και ευχόμαστε να είναι η απαρχή άλλων συναντήσεων που θα διοργανώσουμε με εκπροσώπους της χώρας σας. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την παρουσία σας και για την παρουσία της αντιπροσωπείας σας και ελπίζουμε ότι θα παραμείνετε στις Βρυξέλλες για λίγες ε, ημέρες και ότι η παρουσία σας θα είναι καρποφόρα. Όταν εγώ μίλησα για τον κύριο Μπέλτερ, είπα ε, ότι είναι Ολλανδός και όχι Ισραηλινός, όπως ελέγχθη, και είναι πρόεδρος της αντιπροσωπείας των σχέσεων με το Ισραήλ και συντάκτης μιας γνωμοδότησης που αφορούν τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ιράκ. Και υπέβαλε ένα ερώτημα για την επιρροή του Ιράκ, στον, του Ιράν, στην, στον γεωγραφικό αυτό χώρο. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και χαίρομαι γιατί βρεθήκατε εδώ.